Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στα δοσία σας, στους φακέλους σας. Εάν δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς ε, αλλαγές. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες και της Επιτροπής ΕΝΒΕ και της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Καλωσόρισαν όλοι οι συνάδελφοι των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που εργάζονται από κοινού για να εκπονήσουν αυτήν την σημαντικότατη έκθεση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την ε, πολύ καλή συμμετοχή όσων ασχολούνται με τη σύνταξη της έκθεσης και τη διοργάνωση των εργασιών μας, ιδίως σε ό,τι αφορά την δική μου σχέση συνεργασίας με τον ε, κύριο Γκρότε που είναι και εισηγητής. Οι κοινέ συνεδριάσεις, όπως θα γνωρίζετε, οργανώνονται πάντοτε με την παρουσία την ταυτόχρονη παρουσία των δύο Προέδρων και των δύο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και προκειμένου να διευκολυνθεί ο τρόπος εργασίας μας, έχουμε συμφωνήσει να προεδρεύει εναλλάξ ο κάθε πρόεδρος της Επιτροπής. Η προηγούμενη συνεδρίαση είχε πρόεδρο τον κύριο Γκρότε, σήμερα θα προεδρεύσω εγώ και... και... Ε, Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, και πριν δώσω το λόγο. Για να ξεκινήσει η συζήτηση για τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης, θα έλεγα να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 26ης Σεπτεμβρίου. Και αυτά βρίσκονται στους φακέλους σας. Εάν ούτε εδώ έχετε σχόλια να κάνετε, θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο Γκρότε, εφόσον θέλει να παρέμβει, πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Όντως η συνεργασία μας λειτουργήσε καλά την προηγούμενη φορά. Ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσει να συνεχιστεί και ότι θα καταλήξουμε στους αναγκαίους συμβιβασμού για να, συμβασμού, συγγνώμη, για να έχουμε θέση του Κοινοβουλίου. Γιατί στο πρώτο εξάμεινο του 2014 το Κοινοβούλιο πρέπει να εμφανιστεί και ε, στα μάτια της κοινή γνώμης σαν, σαν το θεσμικό εκείνο όργανο το οποίο συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις. Και επίσης να εμφανιστούμε και να γίνουμε αντιληπτοί ως τέτοιο θεσμικό όργανο στην ε, περίοδο πριν από τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αποτελούμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Γκρότε, ευχαριστούμε πρόεδρε. Ξεκινούμε τώρα τις συζητήσεις μας. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα δίωρο για την όλη συζήτηση. Δέκα λεπτά ένα κεφαλή για τους δύο εισηγητές. Πέντε λεπτά για τον κάθε σκιώδη εισηγητή. Στη συνέχεια δύο λεπτά για τους υπόλοιπους που θα θελήσουν να παρέμβουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντελβό της ΕΝΒΗ για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα γνωρίζετε όλοι το σχέδιο έκθεση που εγώ και ο κ. Σιμάνσκι έχουμε πονήσει από κοινού ω ε, κοινοί θα σα θυμίσω ότι βάσει του άρθρου 51 προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Πρόκειται για ένα συμβαστικό κείμενο που σήμερα ε, μπορείτε να το τροπολογήσετε έως τις 12 Νοεμβρίου. Ε, ένα κείμενο για το οποίο και εγώ ίδια έχω αποβάλει τροπολογίες και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό απαντά σε πέντε βασικές προκλήσεις κατά την απόψη μου. Πρώτον, πώς να επιτύχουμε με τρόπο οικονομικός εφικτό το στόχο των οικονομιών μας και του περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, έπειτα πώ να αποφεληθούμε στο μέγιστο βαθμό από τις ευκαιρίε που προσφέρονται από την πρόκληση αυτή ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που να μην μεταφερθούν εκτός Ευρώπης, ώστε να μην χάσουμε οικονομική δραστηριότητα από την Υπηρώ μας. Τρίτον, πώς να ανταποκριθούμε στι κλιματικές αλλαγές βάσει των ε, νέων τεχνολογικών εξελίξεων και των απαιτήσεων ανταγωνιστικότητα και τη τεχνολογική πρόοδου. Τέσσερα, πώ να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια σε σχέση με τι χώρε εξαγωγή, ε, προκειμένου να υποφεληθούμε και πλήρω από το δικό μα δυναμικό προ του ε, πόρου ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Και τέλο, πώς να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις μας, τις εταιρείες μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες από καλύτερες τιμές της ενέργειας για να μπορέσει να ενισχυθεί η αγοραστική τους δύναμη και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να βεβαιωθούμε ότι το κόστο είναι στο δυνατόν χαμηλότερο, αλλά και το κέρδο είναι στο δυνατόν μεγαλύτερο. Αυτό θα μπορέσει να δώσει ένα σαφέ μήνυμα, ένα μήνυμα τελείω σαφέ από την πλευρά του Κοινοβουλίου και μετά την δημοσίευση της Λευκής Βεβλίου της Επιτροπής τον περασμένο Ιανουάριο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου της περασμένης χρονιάς. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή θεώρηση, όσο δυνατόν ακριβέστερη και πιο ε, λεπτομερή για το πώς έχει κατάσταση σε σχέση με το κλίμα αυτή τη στιγμή, ποια είναι η δική μας η δυνατή συμβολή και ποιοι οι στόχοι μας. Η δέσμη μέτρων για το κλίμα λοιπόν, ε, το είχαμε πει και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, έχει να κάνει περισσότερο με τις πολιτικές εθνικών επιδοτήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κάποιες χώρες έχουν αποφασίσει να στηρίξουν και επενδύουν ε, τα μέγιστα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την διάσταση τη αποτελεσματικότητα του κόστου και τη ε, κερδοφορία. Εδώ λοιπόν κάποιε από αυτέ τι ανανεώσιμε τεχνολογικέ λύσει έχουν ήδη οριμάσει και παρόλα αυτά επιδοτούνται ακόμη πολύ εντατικά, ε, προκαλώντα τρέβλωση στην υπόλοιπη ενεργειακή αγορά. Λόγω χάρη στη δική μα χώρα με το φυσικό αέριο. Μια, χώρα, μια, πηγή ενέργεια που ε, ρηπαίνει αρκετά και θα μπορούσε να είναι μια συμπληρωματική λύση σε σχέση με τι ανανεώσιμε πηγέ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε καταχρήσει ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάποιες υπερβολές, με μια σχετική τεχνολογική ουδετερότητα θα έλεγα σήμερα ως προς αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να δεχόμαστε τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, χωρίς καμία αντίρρηση. Δεν θα έπρεπε, να αμφισβητήσουμε την νομιμότητα των στόχων των ανανεώσιμων βεβαίω, γιατί οι εθνικέ πολιτικέ στήριξη ήταν μη αποτελεσματικέ. πρέπει να διευκρινίσουμε όλε αυτέ τι πολιτικέ επιδότηση και στήριξη, να γίνουν πιο συνεκτικέ και να σκεφτούμε εάν ενδεχομένω θα πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη συνέπεια από τα κράτη-μέλη που κάποιε φορέ επιδοτούν ε, και τα ορυκτά καύσιμα πολύ εντατικά. Ε, κατά τα άλλα, ω προ στη δέσμη μέτρων για το κλίμα θα πρέπει να δούμε την επικάλυψη τριών στόχων. Τα αέρια θερμοκηπίου, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την τιμή τη ενέργεια. Κάποιε φορέ υπάρχουν αντίθετε συνέπειε από τι επιδιωκόμενε. Οπότε θέλουμε στην δική μα μελέτη αυτή τη στιγμή, στη συζήτησή μα, να λάβουμε υπόψη τον αλληλοσυσχετισμό μεταξύ των, της πραγματικότητας και των πραγματικών δεδομένων, βλέποντας ότι υπάρχουν συνδυαζόμενα αποτελέσματα μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για το πακέτο του κλίματος πρέπει να αναζητήσουμε ε, το δυναμικό που έχει υποτιμηθεί, αυτό νομίζω θα το εντοπίσουμε με κατάλληλο τρόπο με τους εισηγητές, και αυτό το δυναμικό θα πρέπει να γίνει ένα σημαντικό στοιχείο του μελλοντικού πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια. Τέλος, η ανταγωνιστικότητα, καθώς και όλες οι πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας, είναι στοιχεία που έχουν υποτιμηθεί, για να μην πω ότι έχουν παραγνωριστεί πλήρως ε, ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο που ετοιμάσαμε. Πλαίσιο που αν δεν ε, ενίσχυσε παρκώ την δυνατότητα των κρατών μελών να αποφεληθούν ε, όσο το δυνατόν περισσότερο από τι βέλτιστε πρακτικέ λόγω χάρη που δεν ανταλλάσσονται παρκώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι πλαίσιο θέλουμε να δημιουργήσουμε στο 2030 και σήμερα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, οι εταιρείε, όλο ο μηχανικός κλάδο, οι επενδυτέ αναμένουν αξιόπιστε, σταθερέ, σαφεί απαντήσει με διορατικότητα σχεδιασμένε όχι διαρκείς ρυθμιστικές αλλαγές, ούτε άκερες, διότι δεν μπορούν έτσι να έχουν βεβαιότητα για το τι θα αποφασίσει η Ευρώπη και ότι αυτό θα διατηρηθεί, θα κρατήσει. Ε, διαρκώς αλλάζουμε ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό βεβαίως ε, δημιουργεί ανασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να σβήσουμε από το χάρτη όλα όσα έχουμε δημιουργήσει ως τώρα, για ποιο λόγο. Ο τομέας για τα αέρια του θερμοκηπίου ε, έχει αναπτύξει θέσεις ε, απασχόλησης και είναι πιο αποτελεσματικός από, τα αέρια του από την αντιμετώπιση ε, των κλιματικών αλλαγών με άλλο ε, τρόπο. Ένα εκατομμύρια 200.000 θέσεις δημιουργήθηκαν χάρη στη βιομηχανία αυτή των αερίων του θερμοκηπίου. Αύξηση 3% από το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο αριθμό αυτός θα μπορούσε να ανέβει και να φτάσει τα 3.400.000 έως το 2030 με τις απαραίτητες επενδύσεις, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν. Είμαι λοιπόν υπέρ σε ένα πλαίσιο που να βασίζεται σε τρεις δεσμευτικούς στόχους. Προσέξτε το αυτό. Τρεις δεσμευτικούς στόχους, ναι, αλλά με πολυάριθμες διορθώσεις ώστε το σύστημα να γίνει εύρυθμο και να καταργηθούν οι ασυνέπειες. Τρία στόχοι λοιπόν, αέρα του θερμοκηπίου, ανανεώσιμα και ενεργειακή αποδοτικότητα, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ανταγωνιστικότητά μας, διότι υπάρχει τεράστιο οικονομικό δυναμικό εδώ, και τεχνολογικό και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, παρά τη διάσταση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των εταιριών μας, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στις ε, κλιματικές μας πολιτικές και ενεργικές πολιτικές θα πρέπει να ενσωματωθεί ως ε, έναν απόσπαστο μέρος το κριτήριο του περιβαλλοντικού δυναμικού. Θα πρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένου δείκτες που να επιτρέπουν να μετρήσουμε με σαφήνεια τον αντίκτυπο των επιλογών που γίνονται ως προς την ανταγωνιστικότητα. Πέραν των στόχων μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που λέω ναι στις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, το έχετε καταλάβει προφανώς, και μέχρι να δούμε τι γίνεται με μερικέ άδειε, όπω τη Γερμανία. Ε, γιατί κάποιε χώρε έχουν ε, αυξήσει πολύ γρήγορα τι δυνατότητε παραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Παρόλα αυτά, ε, παραμένουν μέρο τη λύση οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αναπόσπαστο. Και βεβαίω θα πρέπει να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα και να δούμε τι εθνικέ πολιτικέ στήριξη, όπω είπα πριν. Αλλά δυο φορέ ναι στην ενεργειακή αποδοτικότητα, διότι τη αξίζει να είναι ο ακρογωνιαίο λίθο τη κλιματική μα πολιτική και τη ενεργειακή μα πολιτική. Απλώ λίγου αριθμού. Ξέρουμε ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγέα ε, ενέργεια στον κόσμο. Από το 2001 ο λογαριασμό τη ενέργεια τριπλασιάστηκε για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 θα εισάγει το μεγαλύτερο μέρο του πετρελαίου τη και το 83% του αερίου τη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να μην παραβλέπουμε αυτά τα στοιχεία γιατί η... είναι 10% ετησίω η αύξηση του παγκόσμιου αγορά για την ενέργεια και αποδοτικότητα. Εάν δείτε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρέπει να πετύχουμε το 1% τη ενεργειακή αποδοτικότητα μέχρι το 2020 με οικονομία χιλίων εργοστασίων άνθρακα ή ακόμα περισσότερων που κινούνται με πετρέλαιο. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταργήσουμε την ασυνέπεια και να βελτιώσουμε τη συνεργασία, την ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ε, και σε επίπεδο ε, διακρατικό και μεταξύ των εθνικών δικτύων. Ένα παράδειγμα εδώ. Οι χώρες της Μπενελούξ, η Γερμανία και η Γαλλία από το 2005 δημιούργησαν το φόρουμ, το πολυμερές φόρουμ για την ενέργεια. Μιλάμε για ένα φόρουμ ε, προτεραιότητας για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των φορέων, όλων των υπευθύνων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό, κάτι που επιτρέπει να δημιουργηθεί μια τοπική ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Γιατί λοιπόν να μην δημιουργήσουμε βάση τέτοιων προτύπων και άλλα τέτοια φόρουμ ώστε να ε, βελτιωθεί η δυνατότητα διασύνδεση των κρατών μελών. Αυτό δεν θα πρέπει να μα εμποδίσει βεβαίω να μελετήσουμε και την περίπτωση να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη ε, ούτως ή άλλως συνομιλούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να λάβουν ενεργειακές ή κλιματικές αποφάσεις ε, εφόσον μπορεί να επηρεάζουν και τα όμορα κράτη. Και δύο λόγια για το σύστημα ανταλλαγής ε, δικαιωμάτων. Για να αποφύγουμε στο μέλλον one-shot μέτρα όπως το backloading ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και να σταθεροποιήσουμε την τιμή του άνθρακα. Να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα διόρθωσης το οποίο να λαμβάνει υπόψη το οικονομικό πλαίσιο και το πώς προχωρούν οι πρωτοβουλίες μας για τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, λίγα λόγια ακόμη, γιατί δεν σχολίασα, δεν το συζητήσαμε, για το επίπεδο φιλοδοξιών που θέλουμε να ορίσουμε για τους στόχους μας. Δεν το έκανα αυτό και Πραγματικά είναι κάθε φορά πόλεμο οι αριθμοί σε τέτοιου είδου εκθέσει, αλλά για μια φορά θα θέλω τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσοστά, να μην, να μην αποκρύψουν μάλλον τη δυνατότητα να υπάρχει ένα σαφέ μήνυμα επί τη ουσία ω προ το επίπεδο των φιλοδοξιών μα και των στατικικού μα στόχου. Αυτό νομίζω ότι είναι το στοιχείο προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ντελβό. Και τώρα ο κύριο Σιμάνσκι. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη με τα όσα εξήγησε η συνάδελφός μου έχουμε καλύτερη εικόνα. Μαζί με την κυρία Ντελβό μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Και τους δύο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προχωρήσουμε σε μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα χωρίς ωστόσο να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η οικονομία. Και οι δύο επίσης ενδιαφερόμαστε να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης στη βιομηχανία. Πρέπει να προστατευτεί η απασχόληση. Και μας απασχολεί και τους δυο το ίδιο η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας και η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγόμενες μόρφες ενέργειας. Και βεβαίως να διατηρηθούν και καλές τιμές ενέργειας για να μπορέσει να παραμείνει η οικονομία ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι πώς συνδυάζονται αυτά. Είμαι βέβαιος ότι για να περάσουμε σε οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα δεν θα μπορέσει να γίνει εάν δεν αναλύσουμε σε βάθος τις τρέχουσες πολιτικές. Πρέπει να θέσουμε τις εξής ερωτήσεις. Είναι αποτελεσματικό από άποψη κόστου να υποχρεώνουμε τρεις φορές τις ίδιες επιχειρήσεις ή και τις ίδιες χώρες να κάνουν τα ίδια πράγματα όσον αφορά την απασχόληση, τη δημιουργία απασχόλησης, είναι πολύ εύκολο να λέει κανείς λόγια για την αξία των συνδικάτων και για τους πολίτες, για τις πράσινες ε, θέσεις εργασίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Αν εξετάσουμε τις στατιστικές θα δούμε ότι και οι πιο αισιόδοξε προβλέψεις για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης δεν ανέρχονται σε παραπάνω από 2-3 εκατομμύρια συνολικά θέσεις εργασίας. Όμως η οικονομία, η οικονομία υψηλής έντασης ενέργειας εξασφαλίζει πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και δεν κατανέμονται ίδια σε όλους τους τομείς. Για να μετακινηθούν λοιπόν όλες αυτές οι οικονομίες, ιδίως των νέων χωρών, σε μια οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακος δεν είναι εύκολη γιατί δεν είναι και προετοιμασμένη. Ως Ευρώπη είμαστε περιορισμένοι όσον αφορά την πρόσβαση στο δυναμικό αυτό. Και η αγορά ίδια δεν είναι έτοιμη να υιοθετήσει τις μη συμβατικές πηγές ενέργειας. Ίσως μάλιστα αυτό να σημάνει να σημάνει ότι κάποτε μπορεί να μειωθούν και οι τιμές ε, του πετρελαίου. Χρειάζεται συνδυασμός πολλών πολιτικών εάν θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να στοχεύσουμε στην πολιτική του κλίματος έτσι ώστε να απηχεί την κατάσταση των οικονομιών μας. Όχι όλου του κόσμου, της Ευρώπης. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι είδους επιβαρύνσεις έχουν χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, οι Ενωμένε Πολιτείε. Γιατί έχουμε συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές ή θα έχουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα αυτά ευρύτερα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δικό μας μερίδιο <clears throat> της ρήπανση από διοξίδιο του άνθρακος της παγκόσμιας ατμόσφαιρας είναι πολύ περιορισμένο και θα μειωθεί και άλλο. Ας λησμονήσουμε λοιπόν αυτή την ιδέα ότι δήθεν η Ευρώπη μόνη της μπορεί να ρυθμίσει το πρόβλημα του κλίματος. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το πολιτικό δυναμικό που διαθέτουμε για να δώσουμε παράδειγμα. Είπα και στην αρχή ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε παράδειγμα με τις πολιτικές που ακολουθούμε, διότι ελπίζουμε ότι η επιτυχία την οποία μπορεί να καταλήξει η πολιτική προστασία του κλίματος που θα ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα για άλλους. Για την ώρα όμως κανείς δεν προσπαθεί να ακολουθήσει τα βήματά μας. Και γι' αυτό κανείς δεν είναι ικανοποιημένο από το status quo, διότι η πολιτική αυτή δεν έχει αποδώσει, δεν έχει ικανοποίησει τις προσδοκίες. Χρειαζόμαστε και ένα σύνολο κανόνων, διότι για την ώρα δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες για τους επενδυτές στην Ευρώπη. Δεν είναι βεβαίως μόνο ο μόνος φταίχτης η περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές οι οποίες εν τέλει κάνουν πολύ δύσκολο να επενδύσουν οι επενδυτές στην Ευρώπη, διότι αλλάζουν και οι κανόνες. Συχνά πρέπει να φροντίσουμε ώστε η πολιτική κλίματος να πάψει να αποθαρρύνει τους επενδυτές οι οποίοι δεν ξέρουν πώς θα αλλάξουν οι τιμές, είναι άραγε αποδοτικό το να επενδύσουν στην ενέργεια ή όχι. Υπάρχουν πολλοί κακά παραδείγματα και στο παρελθόν όταν έγινε προσπάθεια να αλλάξουν οι κανόνες στη μέση του παιχνιδιού. Για παράδειγμα με το σύστημα ETS, εμπορίας των ε, εκπομπών. έγιναν ριζοσπαστικές αλλαγές πολιτικής και μάλιστα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Και αυτό ήταν πολύ άσχημο για τους επενδυτές οι οποίοι είχαν εμπιστευτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν επενδύσει τα χρήματά τους και εν μια νυχτή έχασαν πολλά. Επαναλαμβάνω ότι η πολιτική για το κλίμα δεν είναι η μοναδική υπεύθυνη, είναι όμως ένας παράγοντας που οδήγησε τι τιμέ ενέργειας στην Ευρώπη να ανέλθουν πολύ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όχι μόνο για τους πολίτες και για τους ε, επιχειρηματίες. Η Ευρώπη δεν είναι κανένα απομονωμένο νησί. Είμαστε μια ήπειρο. Με ισχυρό εμπορικό δυναμικό. Εκπεξεργαζόμαστε τώρα νέες εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά, με τις ΗΠΑ, με την Κορέα και με τις τιμές ενέργειας που διαθέτουμε τώρα είναι αδύνατον. Διότι η οικονομία μας επιβαρύνεται. Και θα επιβαρυνθεί περισσότερο όταν θα εκτεθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, κάτι το οποίο θα γίνει αργά ή γρήγορα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα στρατηγικό στόχο για ένα νέο άνοιγμα της κλιματικής πολιτικής με μια αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στους διάφορους στόχους αηφορίας, ανταγωνιστικότητας, και για μένα ο τρίτος στόχος πρέπει να είναι αυτός της ασφάλειας προμήθειας της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά την, με την κατάσταση βιομηχανιών, βιομηχανιών έντασης ενέργειας. Χρειάζεται να γίνει προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας και ιδίω μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου εμπορίου και να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό που διαθέτει η ενιαία αγορά προς το σκοπό αυτό. Χρειαζόμαστε πραγματικά μια ενιαία αγορά ενέργειας, διότι αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν σημαίνει μονάχα ορθή εφαρμογή του δικαίου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί το δίκαιο αυτό ακόμη δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του από τις χώρες μέλη. Αλλά χρειάζεται να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και στην ανάπτυξη της υποδομής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε άλλες πηγές ενέργειας. Πρέπει να στοχεύσουμε στο ενεργειακό δυναμικό της Ευρώπης, το οποίο είναι υψηλό αλλά δεν είναι ορθά κατανεμημένο. Τέλος, το δυναμικό των χωρών μελών ποικίλει, είναι πολύ διαφορετικό. Εξαρτάται από την γεωγραφική τους θέση, το κλίμα τους, τις εμπορικές και γεωπολιτικές τους σχέσεις κλπ. Όλες οι χώρες λοιπόν είναι πολύ διαφορετικές. Είναι μια... Βρισκόμαστε σε μια ήπειρο, ζούμε σε μια ήπειρο που γνωρίζει πολλές και ποικίλε μορφές. δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στο ΑΕΠ που είναι τόσο σημαντικό για όλους τους πολιτικούς. Πρέπει να δούμε και τις εκπομπές ε, διοξιδίων ή τέλο πάντων ε, αερίων του θερμοκηπίου κατά κεφαλήν και την πορεία από το 1990 και μετά και ποιο είναι το δυναμικό της κινητοποίησης των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας σε κάθε αγορά, κάθε χώρας μέλους και να εξετάσουμε και την αποδοτικότητα της ενέργειας. Οι στόχοι τώρα, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Διότι σε αυτούς πρέπει να καταλήξει η συζήτησή μας για την πολιτική κρίματος. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι τρεις κύριοι στόχοι που έχουμε τώρα είναι πλέον σημαντικοί. Πρώτο λοιπόν, χαμηλού κόστους οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Ορισμένες χώρες μέλη έχουν δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άλλες όχι. Ορισμένες έχουν σε ορισμένα τμήματά τους περάσει σε οικονομίες χαμηλού αποτυπώματος ε, διοξιδίου του άνθρακος και άλλες όχι. Αυτό πρέπει να απηχείτε στο νέο πακέτο για το κλίμα, διότι αν δεν το κάνουμε τότε απλά θα επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα. Και βεβαίως κανείς στον κόσμο δεν θα μας ακολουθήσει. Πρώτο λοιπόν, ο στόχος της μείωσης των εκπομπών πρέπει να υλοποιηθεί με δίκαιο τρόπο, με δίκαιη κατανομή βαρών. Αυτό πρέπει να είναι μια βασική αρχή του νέου πακέτου θα πρέπει να συσχετίζεται με τα όσα αποφασίσαμε για το διεθνές επίπεδο και βεβαίως να είναι καλύτερη κατανομή και στο, μέσα στα πλαίσια του ETS. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιμάνσκι. Ο κύριος Γκρότε τώρα θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Έχουμε επισκέπτες σήμερα από τη Βόρεια Αρινανία Βεσφαλία Σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα, αυτό το κρατήδιο είναι η έβδομη οικονομία στην Ευρώπη. Σας εύχομαι το καλό σωρίσατε. Νομίζω ότι πραγματικά επιλέξατε μια θαυμάσια ημέρα για να μας επισκεφτείτε. Αυτή δηλαδή την ημέρα όπου γίνεται η συζήτηση για τους στόχους του 2030. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όρτκης είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής που είναι από την Βουλή του κρατηρίου Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Ωραία. Καλώ ήρθατε λοιπόν από όλου μα και να ξεκινήσει κατευθείαν η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στου σκιώδει εισηγητέ. Ε, ο κύριο Κουέντρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, κύριος ρόλ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, γι' αυτό εγώ τον αντικαθιστώ. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τη θέση της δικιάς μας πολιτικής ομάδας όσον αφορά το πλαίσιο αυτό 2020 και θα επικεντρωθώ στα πιο επίμαχα ζητήματα που είναι οι στόχοι για το 2030. Συμφωνούμε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από τις εμπειρίες μας και έτσι να καταλήγουμε σε συμπεράσματα για το πλαίσιο 2020. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι στόχοι 2020 επικεντρώνονται υπερβολικά πολιτικές σε βάρος της ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχει άμεση εξάρτηση ανάμεσα δηλαδή στην ενεργειακή πολιτική και την κλιματική πολιτική. Και ήρθε η ώρα, κατά τη γνώμη μας, να επιφέρουμε νέα ισορροπία και να λάβουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία. Το πρώτο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η οικονομική ύφεση μακροχρόνια, η οποία περιορίζει τα δημοσιονομικά των χωρών μελών και περιορίζει και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δάνεια. Δεύτερον, η ενεργειακή πίεση είναι η μεγαλύτερη στον αναπτυγμένο κόσμο. Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές του ηλεκτρισμού αυξήθηκαν 14% περίπου για τα νοικοκυριά από το 2010 μέχρι το 2012 και πάνω από 12% για τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το χειρότερο σύμφωνα με τις προβολές που γίνονται, οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μάλιστα ακόμα περισσότερο. Τρίτον, η Ευρώπη ε, είναι το 11% των παγκοσμίων ε, εκπομπών. Αν το συνδυάσουμε αυτό με έλλειψη φιλοδοξίας από τους εταίρους μας και κύριους ανταγωνιστές μας όσον αφορά τη μείωση του διεξουδίου του Αφρικα, αυτό σημαίνει ότι Όλες μας τις προσπάθειες τις κάνουμε εμείς για μια μείωση η οποία τελικά δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Και πολύ πιθανόν δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε μείωση των εκπομπών μας ή ελάχιστη. Εξάλλου θα εξοικονομήσουμε πολύ λιγότερο από άλλες εκπομπές εκτός ε, Ευρώπης. Θυσιάζουμε δηλαδή έτσι τη δικιά μας την βιομηχανία. Έχοντας υπόψη όλα αυτά, καταλήγουμε στο ότι πρέπει να υπάρξει νέα ισορροπία όσον αφορά ε, τη βιωσιμότητα του περιβάλλον και να τη συνδυάσουμε με την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας για το 2020 και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Όσον αφορά τον στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εννοείται δεν έχουμε τίποτα εναντίον τους, αλλά προς το παρόν η επιπτώσεις στην τιμή της ε, ενέργειας είναι μεγάλες. Παίρνουν επιδοτήσεις και το αποτέλεσμα είναι καταστραφικό για ορισμένες χώρες μέλη. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πια αν θέλουμε να στηρίξουμε πάλι τέτοιους δεσμευτικούς στόχους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι παρετούμαστε από τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Όχι τα ταμεία για την έρευνα και την ανάπτυξη θα βοηθήσουν τις ανανόσιμες πηγές για να φτάσουν σε μια τεχνολογική οριμότητα η οποία να τις καταστήσει και ανταγωνιστικές. Δεν μπορούμε αναδρομικά να υιοθετήσουμε μέτρα σε σχέση με τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Ούτε βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε έτσι στα τυφλά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν είναι ακόμα ανταγωνιστικές και δεδομένου ότι δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα η ενσωμάτωσή του στο δίκτυο. Συνεπώς, θέλουμε πιο καθαρή ενέργεια, αλλά να μην βασιζόμαστε τόσο στις ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, θα έπρεπε να δούμε μήπως θα έπρεπε να βάλουμε και έναν υποστόχο που έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση και μήπως έτσι θα μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα να εξοικονομήσουμε χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιστρέψουμε, θα διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν στα πλαίσια του 2020, όπου ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση ήταν ενδεικτικός μόνο, ενώ για τις ανανόσιμες πηγές ήταν δεσμευτικός. Τέλος, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενεργειακή πολιτική και η κλιματική πολιτική είναι δύο πράγματα συνδεδεμένα μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ένα και το αυτό. Οπότε, να συνεχίσουμε τις προσπαθειές μας για μείωση των εκπομπών, όμως χωρίς να πυροβολούμε τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε και τώρα η συνάδελφος Ουλφκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Όμως ο χρόνος περνάει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει σαφή θέση όσον αφορά την ενεργειακή του πολιτική και την πολιτική για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα παρουσιάσουν τη θέση τους στις αρχές της επόμενης χρονιάς και πριν την άνοιξη του 2014. Η μελλοντική λοιπόν πολιτική αυτή θα εξεταστεί στο Αρενό Συμβούλιο. Βέβαια είναι ανησυχητικό το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφωνίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βασική μας θέση. Ο συνάδελφος Βιντάλ Κουάδρας αναφέρθηκε σε αυτά, με τα, αυτά με τα οποία συμφωνούμε. Όμως υπάρχουν και ένα σωρό με τα οποία δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι η βάση του πρώτου αυτού κειμένου που συνέταξαν οι εισηγητές είναι κάπως περίεργο. Αρχίζει από την βασική θέση που λέει ότι η ενεργειακή ιδιωσιμότητα τελικά απειλεί την ανταγωνιστικότητά μας. Εγώ έρχομαι από ένα μέρος της Βόρειας Ευρώπης που είναι ιδιαίτερα βιομηχανικό, εκβιομηχανισμένο. Και ξέρω πώς επηρεάζεται το περιβάλλον. Οπότε για μένα η ανταγωνιστικότητα σημαίνει ενεργειακή βιωσιμότητα και προστασία του κλίματος. Για μένα έτσι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι θα είμαστε στο μέλλον ανταγωνιστικοί. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να αποφεύγουμε, να εφαρμόζουμε, να αναπτύσσουμε συστήματα τα οποία θα επηρεάσουν πάρα πολύ τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο μέλλον. οι κλιματικές μας πολιτικές προς το παρόν είναι επιτυχείς γιατί μειώνονται οι εκπομπές. Συνεπώς δεν πρέπει να καταστρέψουμε την πορεία αυτή ξαφνικά αλλάζοντας ρότα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η οποία δεν έχει καμία σχέση με το κλίμα. Συνεπώς ομολογώ ότι εξεπλάγει που οι συγητές δεν πάνε ακόμα πιο μακριά, τουλάχιστον σε κάποια σημεία. Είναι καλό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα με αυτή την πρώτη έκθεσή μας για το πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή απόδοση και πάρκια. Θα ήθελα μια σαφή πρόταση. Ανταυτού όμως το κείμενο τι λέει. Λέει ότι θέλουμε μια καλύτερη προσέγγιση της Ευρώπης για την ενεργειακή επάρκεια. Εντάξει. Ωραία, ναι, να το κάνουμε. Να σχεδιάσουμε μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση, αντί να λέμε ότι μάλλον τη χρειαζόμαστε. Η δουλειά μας αυτή είναι, να κάνουμε προτάσεις σεβόμενοι την κατάσταση των κρατών μελών βέβαια, αλλά να είμαστε σαφείς πού θέλουμε να φτάσουμε, ποιος είναι ο στόχος μας, αντί να κάνουμε γενικές ε, έτσι, δηλώσεις. Επίσης χρειαζόμαστε νούμερα, επίπεδα για τους νέους στόχους. Τους στόχους για το 2005 όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, 85%. Τους στόχους αυτούς πρέπει να τους θέσουμε σαφώς και να τους έχουμε συμφωνήσει η μείωση διοξιδίου του άνθρακα επίσης, η επέκταση των ανανόσιμων πηγών ενέργειας και η ενεργειακή επάρκεια. Όλοι αυτοί οι στόχοι επίσης πρέπει να είναι δεσμευτικοί, αλλιώς δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Και κάθε χώρα βέβαια θα αποφασίσει πώς θα πετύχει τους στόχους αυτούς. Δεν λέω ότι εμεί πρέπει να πάμε στι χώρε μέλη και να του πούμε εμεί πώ θα πετύχουν του στόχου αυτού, αλλά οι στόχοι πρέπει να τεθούν με σαφήνεια και να είναι δεσμευτικοί, υποχρεωτικοί. Αν δεν ανανεώσουμε και δεν ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες μας, τότε θα δίνουμε την προτεραιότητα στα ορυκτά καύσιμα. Αν δεν είμαστε αρκετά σαφείς, αν ε, κάνουμε γενικές δηλώσεις μόνο στις εκθέσεις που συντάσσουμε, τελικά άλλες προτεραιότητες θα έχουν το πάνω χέρι αναπόφευκτα. Θα είναι πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις που θα πρέπει να κάνουμε αν δεν ενισχύσουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Και τελειώνω με το εξή. Μου λέει ο πρόεδρος ότι πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε πιο ειδικοί και συγκεκριμένοι. Αυτά. Ευχαριστώ. Τόμσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω με την ανταγωνιστικότητα. Όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Βαρόσο, στις 8 Ιανουαρίου του 2007 παρουσίασε τα πρώτα περί στρατηγικής για το 2020. Η επιχειρηματολογία του ήταν η ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στην πράσινη οικονομία και μόνο επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την πράσινη δηλαδή οικονομία, μόνο τότε θα επιβιώσουμε και θα είμαστε πράγματι ανταγωνιστικοί. Συνεπώς, είναι ενδιαφέρον που βλέπουμε σήμερα ότι η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και πολλές άλλες χώρες επενδύουν πολύ περισσότερα στην ε, οικονομία αυτή από ότι εμείς. Δύο μήνες αργότερα είπαμε ότι δεν φτάνει να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, ότι χρειάζονται και επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο και πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς τις επιχειρήσεις. Χωρίς πλαίσιο για επενδύσεις δεν θα έχουμε επενδύσεις. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι αφελείς, που λένε ότι οι επενδύσεις πρέπει να έρχονται από το κράτος. Όχι, όχι από τα κράτη, από ιδιωτικές πηγές πρέπει να έρχονται οι επενδύσεις. Χωρίς εγγύηση όμως, χωρίς πλαίσιο, κανένας δεν θα έρθει να επενδύσει στην πράσινη οικονομία και στην ε, οικονομία της ενέργειας. Οι τιμές τώρα που έχουμε στην Ευρώπη δεν έχουν καμιά σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Οι τιμές εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Το 2010 250 δισεκατομμύρια ε, δαπανίσαμε που είναι το ίδιο ποσό όπως το ετήσιο ΑΕΠ της Πολωνίας. Γι' αυτό και οι τιμές ενέργειας είναι τόσο υψηλές στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, από την εξάρτηση και να διασφαλίσουμε ενεργειακή επάρκεια, να μην εξαρτώμαστε από τον Πούτιν και από άλλα καθεστώτα, Μέσα Ανατολή ή άλλα από όπου προμηθευόμαστε ενέργεια. Αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν θέσουμε στόχους για ενεργειακή επάρκεια. Κάποιες χώρες μέλη το κάνουν και το πετυχαίνουν γιατί έχουν δεσμευτικούς υποχρεωτικούς στόχους για την ενεργειακή επάρκεια και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το κάνουμε και να στείλουμε έτσι ένα μήνυμα προς τις βιομηχανίες ότι μπορούν να επενδύσουν στην ανανεώσιμη ενέργεια και να μην ανησυχούν για τις επενδύσεις τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν δεσμευτικούς στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμψεν. Και τώρα ο κύριος... Η κυρία Γκερμπράντη. Ο κύριος Γκερμπράντη. Να μιλήσω, μάλλον να αφήσουμε τη συνάδελφο να μιλήσει πριν από την προηγούμενα για μέρος των ελευθέρων. Κυρία Χολ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω εγώ στη θέση του συναδέλφου. Ε, είναι πολύ σημαντικά τα σχόλια που ακούσαμε από σήμερα το πρωί ε, και από του δύο συγγητέ για, τη σημαντικότητα της ενεργειακής, για τη σημασία τη ενεργειακή αποδοτικότητα και τον τρόπο να περιοριστεί η χρήση του άνθρακα και από τον κύριο Κουάντρα, ο οποίο ανέφερε την ε, σημασία του συνολικών στόχων για την ενεργειακή υποδοτικότητα. Εύστοχα λοιπόν αυτά τα σχόλια και είναι σημαντικό διότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι προς τη στιγμή, προς στιγμή 60% της μείωσης αερίων του θερμοκοιμίου που κάνουμε ε, και καταφέρνουμε δεν είναι από το σύστημα ανταλλαγής αλλά από την υπόλοιπη το άλλο σκέλος της πολιτικής μας. Αυτό που να τονιστεί λοιπόν στην, αίσθηση, στην έκθεση και σε αυτό να συμφωνήσουμε. Ξέρουμε ότι από την σκοπιά της ενεργής αποκοτικότητας πρέπει να την τονώσουμε και πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να υποβάλουν εκθέσεις και αυτό γίνεται ήδη στα, βάση, στα πλαίσια του οικονομικού εξαμήνου. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια από την πλευρά του εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τιμών της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση, χρήση ενέργειας και εθνικοί φορείς μας είπαν πρόσφατα ότι πρέπει να θεωρεί την ενεργειακή αποδοτικότητα στο πρώτο καύσιμο και η πρωταρχική πηγή του τροφοδότησής μας. Πόση ενεργειακή αποδοτικότητα λοιπόν χρειαζόμαστε από οικονομικής σκοπιάς. Πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπε ένα Ινστιτούτο Μελετών ότι πρέπει να, να βελτιώσουμε κατά 40%. Μπορούμε μάλλον να βελτιώσουμε κατά την 40% την ενεργειακή μας αποδοτικότητα στο 2030. 61% στα κτίρια και 40% στις μεταφορές μπορούμε να έχουμε. Εάν λοιπόν αυτό το οικονομικά ζωτικό στοιχείο της ενεργικής αποδοτικότητας όντως τονιστεί. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το 2030. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πριν θέσουμε τους στόχους για τα αέρια του θερμοκηπίου, διότι στην πράξη βλέπουμε ότι το σκέλος εκτός ETS είναι αυτό που φέρνει ε, την αλλαγή. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου υπάρχουν ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εάν πετύχουμε οικονομικό ωφέλη από την ενεργειακή αποδοτικότητα θα πετύχουμε ταυτόχρονα και τα μείωση των αερίων του ανθρωποκηπίου, πράγμα που ούτως ή άλλως θέλουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σκεφτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε και μετά το 2030. Και φτάνοντας στους ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι έχουν επιτύχει ε, ω τώρα και με το, μέχρι το 2020 θα έχουμε πετύχει ένα μεγάλο μέρο των στόχων μα. Θα, ε, θα έχει αυξηθεί και η ποσότητα των ε, πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε από ανανεώσιμα και το κόστος θα έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά το θέμα είναι εάν έχουμε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση κατά την ύφεση που διανύουμε. Έγινε πολλή συζήτηση τελευταίω και ιδίω σήμερα το πρωί για το κόστος τη ενέργεια. Το κόστος καθώς θα έπρεπε να απομυθοποιήσουμε κάποια στοιχεία που συχνά ε, ακούγονται. Λόγου χάρη, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δεν είναι ο λόγο που αυξήθηκαν οι τιμέ τη ενέργεια. Καθόλου δεν είναι αυτό ο βασικό λόγο. Αυτό το αρνούνται κατηγορηματικά οι ειδικοί. Οι τιμέ ε, του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων φταίνε. Η ενέργεια από τι ανανεώσιμε πηγέ είναι ένα ελάχιστο ποσοστό από τη συνολική κατάσταση που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργεια. Έπειτα, οι επιδοτήσει δεν ε, είναι αποτελεσματικέ. Όχι, είναι, αλλά πρέπει να σχεδιαστούν καλύτερα να είναι καλύτερα στοχευμένε και καλύτερα διορθωμένε. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε προβλήματα για τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι αν δηλαδή συνεχίσουμε να στηρίζουμε τεχνολογίε στη φάση ορίμανση, δημιουργείται πρόβλημα και βεβαίω μένουν μετά και άλλα προβλήματα στην πορεία. Πρέπει να συζητήσουμε το πώ θα επιδοτήσουμε τι ανανέωσιμε πηγές στο μέλλον και να επικεντρωθούμε στι τεχνολογίε σωστή μέτρηση. Το πρώτο, το τρίτο μάλλον στοιχείο είναι ότι τίνουμε να πούμε ότι θέλουμε να είμαστε ενεργειακά αυτάρκης. Να έχουμε εγχώρια παραγωγή ενέργεια με το σχιστολιθικό αέριο λόγω χάρη, που πιστεύουμε ότι θα είναι μια φτηνή απάντηση, όπω έγινε στι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, στην ε, εκλογική μου περιφέρεια, και εφόσον δεν ήμασταν εδώ, μίλησα πολύ με χημικέ βιομηχανίε. Και όλοι μου είπαν ότι αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε το σχεστολιθικό αέριο στην Ευρώπη δεν θα είναι φθηνό όπω στι ΗΠΑ, θα γίνει ανταγωνιστικό μόνο όταν φτάσει και θα φτάσει πολύ γρήγορα τι τιμέ του φυσικού αερίου που γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με την ενεργειακή μα αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είναι η απάντηση που ελπίζουμε το σχεστολιθικό αέριο, είναι ένα μύθο όλο αυτό. Και τέλο την Επιτροπή Βιομηχανίας όπου συμμετέχω. Μιλάμε πάρα πολύ για την ενεργειακή και βιομηχανική μας ε, πολιτική θα πρέπει να μιλήσουμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια Από την σκοπιά της βιομηχανικής πολιτική. 138 χώρε στον κόσμο το κάνουν. Εάν δεν το σκεφτούμε εμεί θα χάσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο ω Ευρωπαϊκή Ένωση στον χώρο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα πλεονεκτήματα ζητήματα του να παίρνει κανεί στι 6 το πρωί το τρένο είναι ότι μέσα. Μάλλον να παίρνει για 6 ώρε τρένο είναι ότι έχει το χρόνο να διαβάσει εφημερίδε. Διάβαζα λοιπόν του New York Times σήμερα το πρωί, τη στήλη του Thomas Friedman και θα σας διαβάσω μία πρόταση. Το θέμα είναι η ρήπανση ατμόσφαιρα στην Κίνα. Λέει λοιπόν, αν η Κίνα ανταποκριθεί σε όλα τα κριτήρια της οικονομικής επιτυχίας εκτός από ένα, του να μην μπορείς να ζήσεις εκεί, τι νόημα έχει. Λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ, γιατί πολύ μου αρέσει όλη αυτή η οικονομική επιχειρηματολογία που αναπτύσσουμε εδώ, αλλά αν με όλα αυτά τελικά δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ, τι νόημα έχει. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο Φρίντμαν, είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους εγώ πιστεύω ότι η Κίνα θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε τώρα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτή η ρήπαση της ατμόσφαιρας έχει να κάνει και με το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν ο Τόμας Φρίντμαν είναι ένας ε, ε, φανατικός του περιβάλλοντος, υπάρχουν και άλλες πηγές. Από το Waterhouse Coopers, λογιστική εταιρεία, που πολύ πρόσφατα είχαν την έκθεσή τους για το 2013 που αναφέρεται στην οικονομία δίκτυ χαμηλού ε, αποτυπώματος άνθρακα. Για το 2008 λοιπόν έχουν υπολογίσει και εδώ δεν μιλάω μόνο για περιβαλλοντολόγους, έτσι, μιλάω για λογιστές που ξέρουν πώς να υπολογίζουν τα πράγματα. Υπολόγισαν λοιπόν ότι για να διατηρηθεί ανάπτυξη χωρίς να ξεπεράσουμε την θέρμανση 2 βαθμούς, τότε θα πρέπει τζοχτό να μειώσουν σε 3,5% το αποτύπωμα άθρα κόστους. Για την ίδια χρονιά, στην έκθεση αυτή δηλαδή, το αναλύσανε και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 3,5% το χρόνο δεν γίνεται, είμαστε στο 0,7%. Και άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο. 6% μείωση αποτυπώματος άνθρακα κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο μέσο όρο αυτό. Busting the Carbon Budget λέγεται η έκθεση αυτή. Γιατί το 34 θα έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το ε, ποσό που έχουμε για τον άνθρακα αυτού του αιώνα. Νομίζω ότι όλα αυτά ξεκαθαρίζουν την κατάσταση. Όμως δεν πρόκειται μόνο για το κλίμα. Δεν μιλάμε μόνο για το κλίμα όσον αφορά το πακέτο αυτό για το 2030. Υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός στόχος κατά τη γνώμη μου και αυτός είναι να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό σε ικανοποιητικές τιμές για την Ευρώπη, για το μέλλον. Η Ευρώπη είναι πολύ ευάλωτη γιατί έχουμε ελάχιστα ορυκτά Άρα έχουμε πολύ λίγες δυνατότητες να έχουμε αυτή την ενεργειακή επάρκεια. Και ακόμα και τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα, εντάξει το του, για το διεξίδιο του άνθρακα από, τη ΣΕΛΟ ο κύριος Φώσερ, λέει ότι ο σχιστόλιθος δεν έχει μέλλον στην Ευρώπη. Και είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει λεφτά από αυτή την υπόθεση. Ε, λοιπόν, αυτός ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει μέλλον για το σχιστολιθικό αέριο. Αν λοιπόν δεν έχουμε ορυκτά ούτε καν ε, τα μη συμβατικά, ε, τότε πώς θα διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό είτε με την πυρηνική ενέργεια είτε με τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Για μένα τα πυρηνικά έχουν τεράστια μειονεκτήματα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά σημαίνει ότι θα εξαρτώμαστε από άλλες περιοχές του κόσμου, όπως ισχύει και τώρα με τα ορυκτά. Συνεπώς πρέπει να επικεντρωθούμε στις ανανεώσιμες, όχι μόνο για λόγους κλίματος, αλλά και εξαιτίας ε, της επιθυμίας μας να έχουμε ενεργειακή επάρκεια με χαμηλό κόστος. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το σφάλμα να επιβραδύνουμε τις ε, νεμογεννήτρες. Όχι, θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκός αυτός ο στόχος μας να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω αυτό να αντικατοπτριστεί και στην έκθεση τελικά. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για το κλίμα. Χρειαζόμαστε περισσότερα από δείκτες για το κλίμα. Είναι ξεκάθαρο. Ένας μόνος ενιαίος στόχος για το διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να βοηθήσει για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν θα μειώσει, δεν θα βοηθήσει μάλλον για την ενεργειακή επάρκεια και το κόστος. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την ευημερία των πολιτών μας, πρόκειται και για την μελλοντική μας οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο σε έναν νέο στόχο διοξιδίου του άνθρακα, αλλά στην ενεργειακή επάρκεια και τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Και ας το δούμε κατάματα. Πού πετυχαίνουμε περισσότερο, στις ανανεώσιμες πηγές, γιατί είναι δεσμευτικός ο στόχος. Άρα για μένα είναι ξεκάθαρο και πάλι χρειαζόμαστε τριπλούς στόχους και πρέπει να είναι δεσμευτικοί, υποχρεωτικοί. Ευχαριστούμε, ο συνάδελφος Έγκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους εισηγητές για το πρώτο σχέδιο της έκθεσης που ετοίμασαν. Δείχνει με σαφήνεια που θα μπορούσαν να συγκλίνουν οι απόψει μας. Ε, ε, αυτό ήδη φαίνεται όταν συνεργάζονται δύο συνεισηγητές. Είναι μια ωραία λοιπόν αρχή να ξέρουμε ότι μπορεί και να συμφωνήσουμε. Αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Από την πλευρά των πρασίνων λοιπόν θα σας διευκολύνουμε και θα βελτιώσουμε την έκθεση. Ας το πω έτσι. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν τις δικές μας παρεμβάσεις ως μη βελτίωση, εμείς έτσι τις βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα κάποια σχόλια για το λόγο για τον οποίο συζητάμε έτσι κι αλλιώ για το 2030. Γιατί συζητάμε για το 2030. Είπε ο συνάδελφος μου πρέπει να βασιστούμε σε δεδομένα. Θα συμφωνήσω και έχω δει και εγώ πολλέ από τι μελέτε. Ένα παράδειγμα είναι η μελέτη του IPCC που λέει ότι εκατοντάδε επιστήμονες ε, λένε ότι το κλίμα αλλάζει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνούμαστε το τι συμβαίνει και ας βασιστούμε στα δεδομένα και ας αφήσουμε τις φαντασιώσεις περί κλίματος. Εάν δείτε με προσοχή την έκθεση του IPCC θα καταλάβετε ότι αυτό, που είναι, αυτό που είναι σημαντικό είναι η σόρευση των εκπομπών. Αυτό ισχύει πιο πολύ για το διοξείδιο του άνθρακα. Αν ξεπεράσουμε το 1-3 τόνων ε, διοξιδίου, ξεπερνάμε το 2% του στόχου. Είμαστε ήδη στα μισά του δρόμου. Οι εταιρείε πιστεύουν ότι σε 30 χρόνια θα έχουμε περάσει το 1-3 και πρέπει να δράσουμε, πρέπει να δράσουμε τώρα με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα ως το 2020. Ο δεύτερος λόγος είναι η επενδυτική ασφάλεια. Όλοι οι άνθρωποι που μιλούν εκ μέρους των εταιριών και της βιομηχανίας λένε ότι ένα πράγμα χρειάζεται ο κλάδος, την επενδυτική ασφάλεια. Θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει μετά το 2020. Το 2020 είναι αύριο. Θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει μεθαύριο. Μετά το 2020, δηλαδή το 2030. Επίσης, αυτό το συζητάμε και για σκοπούς διεθνών διαπραγματεύσεων, διότι το 2015 πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Εάν η Ευρώπη φέτος δεν καταλήξει σε ε, στις αρχές της επόμενης χρονιάς, με μια συμφωνία για το τι εμείς υποστηρίζουμε, ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μετά δεν θα μπορέσει να συζητηθεί καμία πρόταση. Πρέπει λοιπόν κάποιος ημεθετηρίας να ε, βρεθεί ώστε να αποφύγουμε τις αποτυχίες τύπου Κομμαχάγης. Επίσης για το επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Πολύ σαφώς, εάν δείτε τι γίνεται με την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή οδεύει στην κατεύθυνση της μείωσης του 30% στο 2020. Είμαστε ήδη πέρα από το 20%. Έχουμε ξεπεράσει με τις μελέτες και τα στοιχεία τον στόχο και οδεύουμε προς το 30% χωρίς προσθήκες, χωρίς ε, εντατικοποίηση. Γιατί λοιπόν να μην φτάσουμε για, το, γιατί να φτάσουμε στο 30% το, το το 2050 μπορούμε να πετύχει το 80% με το 90%. Δείτε τι λένε οι εκθέσεις, δείτε ποιες είναι οι βασικότερες ε, δεσμεύσεις που αυτή τη στιγμή συζητιόνται. 30% έως το 2030. Είμαστε πολύ, στα μισά του στόχου το 2%. Γι' αυτό λοιπόν ας κοιτάξουμε καλύτερα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Λοιπόν, το επίπεδο φιλοδοξιών θα πρέπει να είναι 60% για το 2030. 60%. Τι μορφή θα πρέπει να έχει το υπόλοιπο πακέτο. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για ελεύθερου ή δεσμευτικού στόχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να πάει παραπάνω από το 30%. Λένε ότι θα πάνε στο 50%. Καλό είναι αυτό, δεν είναι πολύ, αλλά καλό είναι. Λίγη περισσότερη φιλοδοξία δεν βλάπτει. Επίση λένε ότι είναι υπέρ όμω των ελεύθερων στόχων. Γιατί ενώ από τη μια υποδιώκουν ένα στόχο, ταυτόχρονα πληρώνουν κατά για την πυρηνική ενέργεια για 40 χρόνια. Και αυτή τη Δευτέρα έμαθα ότι ο κύριος Ντέιβις από το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει και ένα στόχο για το ACCS. Αυτό σημαίνει ενεργειακό πακέτο για το Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο για το διοξείδιο του άνθρακα, άλλον για την πυρηνική και άλλο για το CCS. Ωραία, πολιτική απόφαση είναι αυτό, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε άλλους στόχους για το διοξείδιο του άνθρακα. Εγώ θα προτιμούσα τις ανανεώσιμες πηγές, ας πούμε, όχι το ε, CCS και την πυρηνική. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε συγκεκριμένε πολιτικέ αποφάσει. Και για τι ανανεώσιμε πηγέ, πολύ σύντομα. Μα ε, μας λέει ο κόσμο ότι στρεβλώνεται η αγορά από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό είναι δήλωση των 10 μεγαλύτερων γενικών διευθυντών. Αυτοί το λένε. Διότι το 50% των γερμανικών ανανεώσιμων έχουν φτάσει στα χέρια των πολιτών. Δεν είναι πια στα δικά του χέρια ε, φυσικά τους τρευλώνει τη δική του την αγορά. Δεν τους συμφέρει και εμείς το θέλουμε αυτό. Ναι, δεν θέλουμε την ενέργεια στα χέρια των μεγάλων ε, πολυεθνικών, των 10 μεγάλων πολυεθνικών, στους πολίτες να πάνε. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα των ανανεώσιμων. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν που 10 γενικοί διευθυντές ε, παραπονούνται, αλλά όποιος άλλος τέλος πάντων μπορεί να παραπονιέται, αλλά να, τι πρέπει να κάνουμε για τι ανανεώσιμε και για τι επιδοτήσει. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει το θέμα αυτό. 100 δι ευρώ για τα ορυκτά. 35% μόνο για τι ανανεώσιμε πηγές. Α μιλήσουμε λοιπόν για τις επιδοτήσεις, αλλά ας δούμε καλύτερα πρώτα τα ορυκτά καύσιμα, έτσι. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε επειδή συμφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Ζημάνσκι και ο κύριος Κουάδρας, ε, θα επικεντρωθώ σε μερικά στοιχεία δικά μου, μερικές επισημάνσεις. Η κοινή έκθεση των δύο εισηγητών αποτελεί αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών και θεωρώ ότι θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ακόμα. Πάντως νομίζω ότι η πρώτη παράγραφος στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι μόνο προς το Συμβούλιο. Λέει παράγραφος, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο το Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση για το 2050. Στείλαμε με αυτή την έκθεση ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τα no regrets options τα οποία είναι επιλογές μακροπρόθεσμες με ορίζοντα το 2050. Σε αυτή την έκθεση για το 2030 θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα λύσουμε τα σημερινά προβλήματα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως για παράδειγμα την κατάσταση του ETS και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να μας προβληματίσει το γεγονός ότι και με περισσότερο άνθρακα και ότι η βιομηχανία του φυσικού αερίου βρίσκεται σε κρίση παρόλο που είναι λιγότερο βλαβερό στο περιβάλλον από τον άνθρακα. Επειδή δε πολλά ελέγχθησαν ε, για το θέμα της, ε, των υψηλών τιμών των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να πούμε ότι στην σημερινή κατάσταση δεν μας έφτασε μόνο αυτό, αλλά επίσης και η αναποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων στήριξης των ΑΠΕ και οι υψηλές τιμές βεβαίω των ορυκτών ε, καυσίμων. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε την εικόνα πραγματικά πώς είναι. Σχετικά με τις ΑΠΕ. Ακούω πολλούς συναδέλφους να λένε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ίδια συνταγή δηλαδή business as usual, με νέους στόχους που θα επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με πολύ κόπο στην έκθεση του κυρίου Ρόιλ για τη ΣΑΠΕ. Στην πρώτη παράγραφο του ψηφίσματος καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα πανευρωπαϊκό στόχο για τη ΣΑΠΕ για το 2030. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να θέτουμε ξανά το ίδιο θέμα. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Ρόιλ και για μένα όποιες συζητήσεις γίνονται γύρω από τις ΑΠΕ θα πρέπει να γίνονται με βάση αυτής της έκθεσης. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές επίπεδο, πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθούμε στις εξελίξεις με τις πιθανές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας καθώς και στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή στα ενεργειακά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την προθυμότητά τους να βρουν συμβιβασμούς. Ελπίζω αυτό το πνεύμα να περάσει σε όλους τους κοιόδης και ευελπιστούμε σε επικοδομητικές συζητήσεις στις μεταξύ μας συναντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τζαβέλα. Κλείσαμε με τις παρεμβάσεις των ε, σχεδόν συγητών. Τώρα να ακούσουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία εισηγήτρια καθώς και τον εισηγητή. Συγκαταλέγομαι μεταξύ των ε, προσώπων εκείνων που τάσσονται υπέρ των τριών δεσμευτικών στόχων. Άλλωστε έτσι συζητήσαμε και συνεννοηθήκαμε και στην ε, ομάδα εργασίας για το περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εδώ θέλω να προσθέσω ένα ακόμη επιχείρημα. Στην συνθήκη τη Λισαβόνας λέγεται ότι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να προάγει την, τις ανανεώσιμες ενέργειες. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε και νομικούς που θα μας αποδείξουν ότι μια πολιτική η οποία βασίζεται μονάχα πολιτική ενέργεια, δηλαδή, στον άνθρακα και στην ατομική ενέργεια είναι και παράνομη. Ας μην το λησμονούμε αυτό. Θυμίζω και συμφωνώ με τον Βιντάλ Κουάδρα ότι κάναμε λάθος που δεν καταστήσαμε την αποδοτικότητα της ενέργειας δεσμευτικό στόχο εξ αρχή. Το πιο σημαντικό είναι η καλή απόδοση, η αποδοτικότητα της ενέργειας, διότι και στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα μέχρι τώρα, διότι έτσι μόνο θα μειωθεί το κόστος, διότι και οι επενδύσεις θα αποδώσουν περισσότερο και το συστημικό κόστος θα μειωθεί. Διότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε κάποιο ποσοστό ηλεκτρικού ρεύματος, τότε δεν χρειαζόμαστε ούτε νέες γραμμές μεταφοράς του, σταθμούς, μετασχηματιστές κλπ. Για τους στόχους τώρα θέλω να πω Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια βέβαια. Παρακολουθώ λίγο και τι γίνεται στις συζητήσεις για τη δημιουργία ε, του νέου συνασπισμού στη Γερμανία. Είδα και τι λένε στην Μεγάλη Βρετανία για 40% και για 50%. Η Γερμανία ακόμα απέχει. Σε ένα από τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων λέγεται ότι η γερμανική κυβέρνηση θα ταχθεί υπέρ τουλάχιστον του 40% για το 2030. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι άξιο να υποστηριχτεί και θα κάνω σχετικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίζε. Η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους ε, εισηγητές για την έκθεσή τους. Κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσφέρουμε συνθήκες ασφάλειας για τους οικονομικούς φορείς και κατεπηγόντως να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από το 2020 ε, προς το 2030 και ακόμα πιο μακριά. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να διορθώσουμε κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πακέτο μας για το 2020. Ένα από αυτά τα στοιχεία για τη δέσμη μέτρων είναι ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει και με την ενίσχυση της ιεραρχικής αποδοτικότητας και των τεχνολογικών λύσεων η έρευνα και η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να μειώσουν ε, το κόστο πολλών τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούνται για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στη χώρα μου, λόγω χάρη είναι πολύ σημαντική η ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά. Διότι αν δείτε τι γίνεται με τι υπόλοιπε εταιρείε ανά την Ευρώπη, θα πρέπει και εμεί να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ. Αντιδάλω δεν έχει νόημα εάν δεν έχουμε αρκετά δεν φτάνει. Θέλουμε να μπορούμε να εξάγουμε, να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς ε, συνεργασίας. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο αλληλοσυχητισμός ε, μεταξύ των ε, χωρών, είναι καθοριστικό αυτό. Και για την Παγκόσμια Συμφωνία θα πρέπει η φιλοδοξία των στόχων μας να συσχετιστούν και με την ύπαρξη ή όχι μιας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές. Ως προς την εξισορρόπηση των όσων προβλέπονται ήδη για το 2020. Μια σκέψη. Υπάρχουν πολλές δυνατές ε, περιπτώσεις ή υποθέσεις. Υπάρχουν κάποιες μελέτες πανεπιστημιακές για αυτά και μπορεί να συμβεί. Μπορούμε να έχουμε συνδυασμένου στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αποδοτικότητα αντί να είναι δύο ξεχωριστοί στόχοι. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη. Μπορεί να κάνουν περισσότερα κάποιοι για τις ανανεώσιμες πηγές, ε, κάποιοι μπορεί να κάνουν περισσότερα για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, θα μπορούσαν να το καθορίσουν οι ίδιοι. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο αφετηρίας για να επιδιώξουμε την ασφάλεια μην χάσουμε αυτό ε, στην πορεία, διότι πρέπει ο κλάδος αυτός να γνωρίζει, να καθησυχαστεί. Μια άλλη ιδέα είναι να έχουμε πολιτική ή υποστόχους για την υπερθέρμανση. συμφωνώ και το σύστημα μεταφορών. Συμφωνώ με τη Φιώνα Χόλ Θα πρέπει να είναι ένα συνολικό σύστημα μεταφορών, να χρησιμοποιεί τα βιοκάψιμα, όλες οι ε, προσπάθειες των πόλεων, των αστικών κέντρων, των μεταφορικών δικτύων να ε, ληφθούν υπόψη, ώστε να μειωθεί η ένταση των μεταφορών η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από το απλό πακέτο για το 2020. Δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ε, λεπτομερείς ε, στις λύσεις μας και περίπλοκες στη σκέψη μας για να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Ε, Σημερίζουμε πάντως πολλές από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Λένε. Γιώ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι εισηγήτρια και οι εισηγητής κατέδειξαν τα σημεία εκείνα όπου σημειώνεται συνένεση στο Κοινοβουλίο. Είναι σαφές για όλους μας ότι οφείλουμε να μειώσουμε και άλλο τις εκπομπές. Γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύτιμες πηγές ενέργειας, διότι είναι δικές μας και χρειάζεται να τις διευρύνουμε. Και έχουμε και το θέμα της αποδοτικότητας της ενέργειας, όπου ακόμα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μεγάλο δυναμικό διότι και οι επενδύσεις που θα κάνουμε στον τομέα αυτό θα παραμείνουν στην Ευρώπη. Θα είναι επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και απασχόληση. Αυτά τα τρία θέματα αξίζουν να τα επεξεργαστούμε περισσότερο. Και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω, ότι η έκθεση των δύο εισηγητών είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε πριν καταθέσει προτάσεις η Κομισιόν και έλθει μετά το, την άνοιξη το Συμβούλιο Κορυφής εδώ μπορούμε να πούμε ποια πράγματα θέλουμε για το 2030 και αυτό είναι και η δοκιμασία θάρρους που πρέπει να περάσουμε. Αν όντως δηλαδή μπορούμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Η ενέργεια κοστίζει, είναι ακριβή, σωστό είναι αυτό. Αυτό όμως δεν είναι το φταίξιμο της πολιτικής μας προστασίας του κλίματος. Είναι το αέριο και το πετρέλαιο που είναι ακριβά. Παγκοσμίω δεν έχουν σχέση με τα προγράμματα της Ένωσης. Όποιος λέει ότι η ευθύνη της Ευρώπης είναι μόνο 11% θα σας απαντήσω ότι η Κίνα είναι μεγαλύτερη, ε, στην Κίνα γίνονται οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην αιωλική ενέργεια και οι Κινέζοι είναι αυτοί που προωθούν περισσότερο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει κίνδυνος εκτός των άλλων να χάσουμε και το τρένο της εξέλιξης αυτής. Θα ήθελα να πω στον ε, εισηγητή κ. Σιμάνσκι ότι έχει καλώ στο πακέτο του 2020 έχουμε κατανομή βαρών. Δεν μπορούν να αποδώσουν όλες οι χώρες το ίδιο. Χρειαζόμαστε στόχο συνολικό τη Ένωση, αλλά κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα στις 27 χώρες τότε, 28 νυν, για το ποιο μπορεί να κάνει τι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να επαρεχόμασταν στις απαρχές της πρότασης, της όλης συζήτησης, διότι ίσως κάπου έχουμε ξεφύγει ε, στην πορεία. Οι εκπομπές του δεξιδιού του άνθρακα είναι το βασικό πρόβλημα να μην ε, χάσουμε από τη σκέψη μας αυτό που μόλις είπαν οι συνάδελφοι από τους ε, πρασίνους. Δεν έχουμε μπροστά μας μια γυάλινη σφαίρα. Πολύ σύντομα θα βρεθούμε στη Σύνοδο Κορυφής της ε, Βαρσοβίας και θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Η έκθεση της αίτησης νομίζω δίνει υπερβολική έμφαση στον αντίκτυπο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ίσως λοιπόν να παίξω εδώ λίγο το ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου. Α υποθέσουμε ότι η έκθεση αυτή έχει δίκιο και ότι το 2020 έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Τι σημαίνει όμω αυτό διεθνώ. Ούτε 1% δεν εκπροσωπεί ο στόχο αυτό. σω η μέρα τη καταστροφή, η μέρα του Αρμαγεδόνα το 2050 όπως μας λένε οι πράσινοι που θα πετύχουμε το 2% υπερθέρμανσης στην παγκόσμια θερμοκρασία, μπορεί να έρθει. Α σκεφτούμε ότι πετυχαίνουμε όμω το σωστό στόχο πέντε μέρε πριν. Δεν θα καταλάβουμε καν τη διαφορά. Νομίζω λοιπόν, και σε αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξω, ότι η σκέψη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, τελικά ίσως να μην έχει και τόσο νόημα όταν σκεφτόμαστε τη διάσταση της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα σωστά τονίστηκε από τον κύριο και διότι το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί στο να συντομότερα. Να πούμε ναι στην καινοτομία, ναι στην υψηλή αποδοτικότητα και στις σχετικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έμπερ. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την κυρία Ντελβό και τον κύριο Σιμάνσκι για την εκθεσή του, που αποτελούν τη βάση επί των οποίων μπορούμε να στηριχτούμε για να συμφωνήσουμε. Αλλά θα θυμίσω και τα όσα είπε προφορικά η κυρία Ντελβό και ο Πέτερ Λίζε. Πρέπει να σκεφτούμε στην Ευρώπη πώ μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχει η αλλαγή αυτή που είναι απαραίτητη για διάφορου λόγου, όχι μόνο για λόγου κλίματο, αλλά και πώ θα κρατήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστική. Έχουμε το πακέτο του 2008 Ορισμένα πράγματα λειτουργήσαν καλά, άλλα λιγότερο και άλλα οφείλουμε να τα επικρίνουμε. Είπαμε, βάλαμε κάποιους στόχους για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορούσαν να ήταν και πιο φιλόδοξοι οι στόχοι, αλλά τέλος πάντων κάτι έγινε. Εκεί όπου είναι το μεγάλο έλλειμμα είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας. Παρόλο που πολλοί οι δήμονες μας λένε ότι μα αυτά είναι και τα φρούτα τα οποία είναι πιο όριμα και πιο χαμηλά στο δέντρο. Δηλαδή θα μπορούσατε να δρέψετε τους καρπούς της αποδοτικότητας ενέργειας πολύ πιο εύκολα. Αυτό το χρωστάμε στους καταναλωτές μας και στην οικονομία. Αφετέρου για τις ανανεώσιμες ενέργειες που διαρκώς εμφανίζονται έχουν δοθεί πολλές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Εγώ κοίταξα λίγο τα νούμερα. Θα σας αναφέρω από την παγκόσμια έκθεση του 2012, παγκόσμια κατάσταση λοιπόν έτσι, η οποία λέει ότι το 2011 αφού σε αυτό το έτος αναφέρεται οι επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα ανήλθαν σημαντικά 13% παραπάνω από το 2010 και το 2011 ανήλθαν σε 523 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβαν τα αρκετά καύσιμα. 88 εκατομμύρια για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Κοιτάξτε τη σχέση. Στη ΔΕ Ευρώπη τα πράγματα έχουν ως εξή. Το 2011 26 εκατομμύρια, συγγνώμη, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, δισεκατομμύρια ε, συν, κάποια εκατομμύρια για την προστασία της υγείας 35 δισεκατομμύρια για, τις, ε, για την ατομική ενέργεια και 30 για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Τώρα, να λέμε όλοι, ή να λένε πολλοί, ότι... Να, να, κοίταξε τις... Ε, Βένερ, έχω τα νούμερα. Δεν είναι δικά μου τα νούμερα αυτά. Ο δικός σου επίτροπος ο Έτιγκερ τα έχει βάλει, τα έχει καταθέσει τα νούμερα αυτά. Μιλούμε για δισεκατομμύρια για όχι για τρει εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να, τα, να λέμε ότι για όλα ευθύνονται ε, οι επιδοτήσει στι ανανεώσιμε ενέργειες. Υπάρχουν ειδικέ καταστάσει, όπω στην Πολωνία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκή πολιτική για επιμέρου τομεί και για επιμέρου χώρε. Όπω είπα πρέπει να δει κανεί τη συνολική εικόνα. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Κοραγιάδης Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα τρει παρατηρήσει. Πρώτον, πριν από 10 χρόνια όλα ήταν προβλέψιμα. Σήμερα τι, τα πάντα είναι απρόβλεπτα. Πέραν του γεγονότος ότι έχουμε σχιστολικό αέριο στις Ηνωμένε Πολιτείες, τελικά ο χάλιβας, ε, ο άνθρακας των Ηνωμένων Πολιτείων έγινε πλέον ανταγωνιστικός για τις ευρωπαϊκές εταιρείες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ε, το αέριο της Ευρώπης αντικαθίσταται από άνθρακα που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πάντα αλλάζουν ταχύτατα. Δεύτερη παρατήρηση. Ανάγκη τεχνολογικής ε, καινοτομίας. Η ιστορία των ανανεώσιμων είναι ιστορία επιτυχίας αλλά μπορούμε να φτάσουμε το 30% και πριν το 2020. Πρόκειται για ιστορία επιτυχία. Γιατί να πάψουμε, γιατί να τη διακόψουμε αυτή την ιστορία επιτυχία. Πρέπει να επιδιώξουμε το 40% στο, το 2030. Αυτό βεβαίω κοστίζει, κοστίζει κιόλα όπω υπόθηκε. Όμω τα πάντα κοστίζουν. Και Υπάρχουν πολλές τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται όπως τα εφηδίκτυα για να λυθούν τα προβλήματα των διακοπών ή το κλειδί του προβλήματος. Η και αποδοτικότητα. Δεν... Μάλλον, έχουμε ως τώρα χρησιμοποιήσει αυτόν τον πολύ ωραίο ε, έβυχο όρο ε, με τρόπο ρητορικό. Θα πρέπει να περάσουμε όμως και στην πραγματικότητα. Ε, και επίσης, το διευρωπαϊκά δίκτυα της ενέργειας. Εάν δεν δημιουργηθεί μια τέτοια αγορά, θα χάσουμε σε όλα τα μέτωπα θα χάσουμε ως προς την αποτελεσματικότητα της αγοράς, ως προς την ε, περιβαλλοντική αηφορία. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε έναν κανονισμό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Όμως από ψυχολογικής ε, σκοπιάς, ε, στο επίπεδο των χωρών, τα πράγματα πάνε χειρότερα από ό,τι πριν από έξι μήνες χρειάζεται να δούμε τι γίνεται με τον ενεργειακό προστατευτισμό. Διότι δεν μπορεί οι χώρε, οι περιοχέ και οι περιφέρειε να υπερασπίζονται τον εθνική του απομόνωση. Είναι σημαντικότατο για τι εταιρείε να υπάρχει σταθερότητα, να, υπάρχει, να υπάρχουν σημάδια σταθεροποίηση για του επενδυτέ. Με το έγγραφο αυτό, πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικό, είναι κέρια σημασία, όμω πρέπει να ε, αρθούν από αυτό οι αμφισημίε. Υπάρχουν κάποιε ασάφειε, δεν έχω τώρα το χρόνο να επιμείνω σε αυτέ, αλλά πρέπει πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σαφέ το κείμενο. Γιατί όσο πιο δυνατόν είναι τα σαφή τα μηνύματα που θα αποστείλουμε, τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα για την αγορά. Ευχαριστούμε η κυρία Κορχόλα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προ... τα συναντήθηκα με τους ε, ψηφοφόρου μου, ή τέλο πάντων ενδυνάμει ψηφοφόρου μου. Είχα μαζί μου μια μεγάλη πέτρα στο μέγεθος του πεπονιού και έλεγα ότι η Ευρώπη προσπαθεί να βγάλει από την πέτρα αυτή κάτι, κάτι που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει λιγάκι το πρόβλημα που έχουμε εμεί. Ότι εμεί δηλαδή προσπαθούμε αυτό, με αυτό κάτι να βγάλουμε, όταν οι άλλοι δεν κάνουν καν αυτό. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι αξιέπαινη και πολύ καλά ισορροπημένη. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι χρειάζονται τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλά καλά σημεία. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει στο δρόμο να πετύχει τους στόχους 2020, ότι δείχνει υπευθυνότητα για τις παγκόσμιες εκπομπές οι οποίες θα μειωθούν. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. 4% ε, το 2030. πρέπει να είμαστε μαζί με αυτούς που εκπέμπουν πολύ από την ίδια πλευρά. Κάτι άλλο πολύ θετικό είναι ότι κάποιες ανανεώσιμες ε, πρέπει να οριμάσουν, να ενηλικιωθούν, εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι άλλες όχι. Νομίζω ναι ότι το θέμα της απόδοσης πράγματι πρέπει να έρχεται από την αγορά και όχι από τις επιδοτήσεις που δίνουμε εμείς. Βέβαια και με το ρηκτά. Δεν πρέπει εμείς με επιδοτήσεις να ενισχύουμε τις ανανεώσιμες, γιατί ουσιαστικά δίνουμε λεφτά για μια τεχνολογία που δεν είναι ανταγωνιστική. Είχα μια τροπολογία στην έκθεση που με την οποία ζητούσα από την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη. Και το βλέπω αυτό εδώ. Οπότε πολύ χαίρομαι. Επίσης το θέμα της διαρροής άνθρακα και αυτό χαίρομαι που βρίσκεται στην έκθεση. Τώρα στην παράγραφο 33 λέμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το επ των ε, χωρών όταν καθορίζουμε στόχους. Μα το ΕΠ πρέπει να το βλέπουμε ως εξής, σαν την μεγαλύτερη απόδοση συνήθως στις χώρες όπου έχουν χαμηλό ΕΠ υπάρχει η δυνατότητα για τέτοιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς. Τι πιο θερμές μου ευχέ για τους διαπραγματευτέ που την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αναλάβουν στη Βαρσοβία την ε, διεξαγωγή τη συζήτηση για τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Δικαιωμάτων μάλλον εκπομπών. Δεν ελπίζω πολλά προσωπικά διότι θα πρέπει να δούμε τι έγινε με τις δηλώσεις του Μπαλί για την κοινή αυτή έστω και διαφοροποιημένη. Δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε προτάσεις που να είναι αποδεκτές τουλάχιστον αρκετά ευρέως. Ε, νομίζω οι στόχοι του 2030 είναι ενδιαφέροντες και να κάνω εδώ κάποια σχόλια. Πρώτον, ο εξορθολογισμός εξορθολογισμός για την μέγιστη δυνατή χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό ήταν απαραίτητο. Έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας και μεταφορών με διαρκή υψηλή ένταση, κάτι σαν ραχοκοκαλιά για την Ευρώπη, που να επιτρέπει να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανανεώσιμε πηγές, διατηρώντας την ε, ενέργεια στη μορφή του ηλεκτρισμού, δηλαδή να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην χρήση. Έπειτα πρέπει να σκεφτούμε εάν στο σύστημα θα καλυφθούν και κάποια άλλα στοιχεία όπως η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές που διατίθενται στην ε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, η βιομάζα, τα κατάλοιπα, τα δασικά ή τα γεωργικά και αυτά να μετατρέπονται σε αέριο προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε ε, κυψέλες ή μπαταρίες υψηλής αποδοτικότητας. Εδώ θα μπορούσαμε σε αυτές τις κυψελίδες ιδίω στην περίπτωση των σταθερών οξυδίων, να αξιοποιήσουμε ό,τι διαθέτουμε, γιατί μπορούμε να έχουμε παραγωγή ενέργεια ηλεκτρική 100%. Μεγάλη αποδοτικότητα λοιπόν ηλεκτρική και με αυτό θα μπορούσαμε να καλύψουμε ανάγκε χαμηλή θερμοκρασία. Υπάρχει μια σειρά από καινοτόμε λύσει που στην ουσία θα μα επέτρεπαν να αποφύγουμε την καύση η καύση είναι ο πρωταρχικός λόγος της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και εν μέρει και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ευχαριστώ. συνάδελφος Βάνμπεργκ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, για κύριε Φαντρέν. Ευχαριστώ και τους δύο σκιώδεις εισηγητές. Ε, έχω να πω τα ε, εκ μέρους τους. Για την έκθεση αυτή θα απογοτεύσω την κυρία Κορόλα γιατί εγώ θα υποβάλω τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για το περιεχόμενο αλλά και για το ύφος κυρία Ντελβό. Είναι λιγάκι χαρακτηριστικό. Λέει ότι όσον αφορά τους στόχους είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνώ και εγώ βέβαια, και θέλω να είναι δεσμευτική. Πώς όμως θα το πετύχουμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, το μέλλον του πλανήτη είναι το μέλλον το δικό τους. Κοιτάμε λοιπόν μακροπρόθεσμα το μέλλον της γης και την υγεία των ανθρώπων και την ποιότητα ζωής. Αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα για μένα. Έπειτα η συζήτηση για το θέμα της τιμολόγησης. Το διαβάζουμε στις εφημερίδες, σε όλη την Ευρώπη γίνεται η συζήτηση, ότι πια η τιμή της ενέργειας έχει φτάσει σε απίστευτα ύψη. Χρειάζεται λοιπόν ένα πλαίσιο για τα ορυκτά καύσιμα, που εξακολουθούν να είναι στην αγορά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πετύχουμε συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι σε συμφωνία μεταξύ μας να πούμε την αλήθεια. Είναι κρίμα που δεν έχουμε τον Επίτροπο για την Ενέργεια, ο οποίο κάνει το αντίθετο. Στην έκθεση που έχει συντάξει λέει ότι τα καύσιμα, τα στερεά, τα ορυκτά, ε, επιδοτούνται περισσότερο από τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι κρίμα, αλλά αυτά βγαίνουν από την υπηρεσία του Επιτρόπου. Εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε κάτι τέτοιο. Τα νούμερα είναι αυτά που είναι. Η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πρέπει να επιδοτούνται. Κυρίως οι πηγές εκείνες ενέργειες οι οποίες μπορούν να μας διασφαλίσουν ένα καλό μέλλον. Τώρα με διάφορους ευρωβουλευτές από το ΕΛΚΑ Ας αποφασίσουμε επιτέλους και μετά να προχωρήσουμε σε πιο καινοτόμες ιδέες για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής κλπ. Ευχαριστούμε η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, οι τρεις στόχοι είναι αναγκαίοι και μπορούν να είναι δεσμευτικοί. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας, δεύτερον ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Είναι κάτι που μπορούμε κάλλιστα να συνδυάσουμε με το κλίμα. Τα νούμερα που έχουμε είναι σαφή. Και η συζήτησή μας, συνάδελφοι, με κάνει κάπως να πιστεύω στη συζήτηση που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το 19ο αιώνα, οι κατασκευαστές των αμαξιδίων με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Μα η... το μέλλον της ενέργειας είναι οι ανανεώσιμες πηγές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι τα ορυκτά. Αυτό εννοείται. Οπότε η συζήτηση εδώ μου θυμίζει συζητήσεις άλλων εποχών. Τώρα δεν μπορεί να αφήσουμε άλλες βιομηχανίες Κίνας και λοιπά να μας ξεπερνάνε. Ή το διαδίκτυο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λοιπά είναι τομείς στους οποίους οι δικές μας επιχειρήσεις θα έπρεπε να έχουν ηγετικό ρόλο. Και βέβαια αυτό δεν θα το πετύχουμε με τους ελάχιστους στόχους που εξετάζουμε τώρα. Άρα υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους που εν μέρη επιτυχάνονται και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Τέλος. Είναι σαφές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ιδιαίτερες καταστάσεις. Πολωνία, για παράδειγμα. Όμως αυτό δεν φτάνει ώστε μια ιδιαίτερη κατάσταση να γίνει και ο γενικός κανόνας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα έχω να πω. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που λένε ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία διασυνοριακή περισσότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, περισσότερες συνέργειες και άρα συνδυασμός δεσμευτικών ε, στόχων. Είναι ζωτική σημασία για να αντικαταστήσουμε την κοινοτική μέθοδο που έχουμε για την ενέργεια. Δεύτερον, ανταγωνιστικότητα. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο θέμα διαφορετικών πηγών και πόρων είναι θέμα γνώσης και επιστημών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην τεχνολογία μας. Συνεπώς θέλω περισσότερη γνώση, IPR, ε, πατέντες στον τομέα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της ενέργειας. Να μην χτίζονται μονάδες με γνώση από αλλού, αλλά από μας, από την Ευρώπη. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για την πρόσθετη αξία που έχει η γνώση. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, η ενεργειακή επάρκεια πρέπει να είναι σημαντική για τη βιομηχανία και να αποτελεί το... αυτό το οποίο μας καθοδηγεί στις αποφάσεις μας. Πάλι εδώ σημασία έχει γνώση. Συνεπώς το κύριο μήνυμα που θα στείλουμε πρέπει να είναι γνώση στην ενέργεια που πρέπει να προωθήσουμε γιατί αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ευρώπης. Και τέλος, επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Χρειαζόμαστε χρήματα και πρέπει να δούμε πολύ καλά τις, τους προμηθευτές μας, προμηθευτές μας ε, ενέργειας, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω. Αν όμως δεν τους έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Και τέλος, μα τέλος, συμφωνούμε με αυτούς που λένε ότι η πρόοδος δεν είναι τα λόγια, αλλά προοδευτική δράση για όλους. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα πετύχουμε κάτι το 2030. Ευχαριστώ. Ρούμπικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Η γενική κατεύθυνση είναι σωστή. Τα προβλήματα σημειώνονται στην μεταποιητική μα στην Ευρώπη. Πρέπει να φροντίσουμε η απασχόληση, η απασχόληση να παραμείνει στην Ευρώπη και ειδήσει να μπορέσουν να καταστούν δυνατές και επενδύσεις. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να περιοριστούμε σε πρώτη ανάγνωση στην παραγωγή ρεύματος και όχι στη μεταποίηση, διότι οι καταναλωτές θα κρίνουν εν τέλει ποια προϊόντα θα αγοραστούν, θα καταναλωθούν στο μέλλον. Και να δούμε ποια προϊόντα παράγονται, κατασκευάζονται χωρίς ε, υψηλό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακος που να παράγεται και αυτά να επωφεληθούν από φορολογικά κίνητρα. Νομίζω ότι οι τρεις στόχοι είναι σημαντικό να υποστηριχτούν, κυρίως δε η αποδοτικότητα, αλλά και η ασφάλεια προμήθειας της ενέργειας, που παίζει σημαντικό ρόλο. Η ενέργεια πρέπει να γίνει φθηνή, να μπορέσει να την πληρώσει κανείς. Και αυτό έχει σχέση και με τις κρατικές επιχορηγήσεις. Χρειάζεται εδώ ωστόσο ένα νέο πλαίσιο το οποίο να επιφέρει μια ισορροπία ανάμεσα στις κλασικές ενέργειες που προέρχονται από ρηχτά καύσιμα και στις ανανεώσιμες ενέργειες. Όλες οι μορφές ενέργειας, ενέργειας, εάν εξετάσουμε, θα δούμε ότι τα κόστη είναι πολύ διαφορετικά για την παραγωγή μέχρι και την τελική αποθήκευση. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε οι νέες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες ενέργειες βέβαια χρειάζονται υποστήριξη ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση των δύο είναι καλά ισορροπημένη και ελπίζω να μην αλλάξουν τον γενικό προσανατολισμό της έκθεσης μετά από τα διάφορα σχόλια που ακούν αλλά και τις τροπολογίες που θα λάβουν. Ελπίζω να μείνει η έκθεση ως έχει. Να μην αλλάξει. Κατανοώ πόσο σημαντική είναι η συζήτηση σήμερα. Και βεβαίως θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες όταν θα μιλήσουμε και για τις πολιτικές μας του κλίματος και της ενέργειας για το μέλλον. Ο κ. Βιδάλ Κουάδρας άρχισε λέγοντας ότι η πολιτική του κλίματος κυριαρχεί και ότι κρίθηκε σημαντικότερη από την πολιτική ενέργειας. Πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Να βρεθούν οι στόχοι αλλά και οι μηχανισμοί για την επίτευξή τους. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους μου είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από τα ίδια. Δηλαδή να επιμείνουμε σε αυτά που διαθέτουμε. Να είναι πιο φιλόδοξοι οι στόχοι μας και να δράσουμε ταχύτερα. Αυτό ίσως είναι μία προσέγγιση. Θα μείνουμε στους τρεις στόχους και πώς διασυνδέονται αυτοί οι στόχοι. Αυτά είναι τα, αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτό νομίζω ότι η στάθμιση των διαφόρων στόχων για κάθε μια χώρα μέλος θα πρέπει να είναι διαφορετική, γιατί υπάρχουν χώρες μέλη όπου μπορούν να επιτύχουν κάποιο στόχο, για παράδειγμα την αποδοτικότητα της ενέργειας, είναι λοιπόν εκεί πολύ ευκολότερο να αποδώσουν και άλλες χώρες μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Αλλά όμως, όσον αφορά τους άλλους στόχους, έχουν άλλη πορεία να κάνουν. Όμως ο γενικός στόχος πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών. Αυτά μπορούν να επιτυχθούν με διάφορους τρόπους και αυτή η ποικιλία προσεγγίσεων πρέπει να τονιστεί. Δεν μπορεί να είναι ενιαίου μεγέθους, one fits all. Και μια φράση τώρα για την συνθήκη της Λισαβόνας. Εκεί μιλήσαμε πολύ για την ασφάλεια προμήθειας της ενέργειας και για το να γίνει η Ευρώπη ανεξάρτητη. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να μην το λησμονούμε. Κυρία Πρόεδρε, λέει ο κ. Λάγκεν, νομίζω ότι το σχέδιο εκθέσεως είναι καλό, είναι μια χρήσιμη βάση. Σηκώνει κάποια ακριβέστερη διατύπωση σε ορισμένα σημεία, αλλά έρχεται και επιβεβαιώνει τους τρεις στόχους και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Βέβαια, ανάμεσα στους τρεις στόχους κάτι έχει αλλάξει και μάλιστα μαζικά. Το θέμα της ασφάλειας της προμήθειας και των τιμών έχουν πλέον πάρει το προβάδισμα απέναντι στην προστασία του κλίματος και αυτό έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας. Εάν δείτε ότι οι τιμές παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ λόγω του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου έχουν ήδη κατέλθει κατά 30% και ότι μεγάλες επιχειρήσεις, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεγάλων βιομηχανικών κλάδων επενδύουν για το λόγο αυτό στις ΗΠΑ, αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις ισορροπιών μεταξύ των ανανεώσιμων ενεργειών. Το γερμανικό μοντέλο αποδεικνύεται ότι δεν είναι καλό της παραγωγής ενέργειας και της διοχέτευσης στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων. Και γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Ο κύριος Ζέιμπερ ανέφερε κάποια συγκριτικά νούμερα. Σε αυτά τα συγκριτικά νούμερα της Κομισιόν περιλαμβάνονται μοναχά οι κρατικές επιδοτήσεις. Στην πραγματικότητα ο γερμανικός νόμος για τη διοχέτευση του, της ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο πληρώνεται από τους καταναλωτές με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και οι επιπτώσεις είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που νομίζουν ορισμένοι εδώ. Η υπερπαραγωγή στη Γερμανία της αιωλικής ενέργειας οδηγεί την Πολωνία και τις κάτω χώρες να λαμβάνουν δωρεάν το πλεονασματικό ρεύμα και ταυτόχρονα ενώ οι τιμές στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 6 λεπτά η κιλοβατόρα, στη, στην Ολλανδία κατέληξαν κατά 5 ε, λεπτά του ευρώ. Και όταν λέει εδώ στην παράγραφο 23 στην έκθεση ότι πρέπει να διασυνδεθούν και τα νησιά στο κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο, τι να πω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στη Μάλτα δεν είναι τόσο σημαντικό να έχουν τους αγωγούς, αλλά να περάσουν από το πετρέλαιο στην αιωλική και στην ηλιακή ενέργεια το ίδιο για την Κύπρο. Έχουμε δηλαδή σε ορισμένε χώρες μέλη πόρους, ενεργειακούς πόρους που μένουν ανεκμετάλλευτοι. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχω ακόμα δύο παρεμβάσει, όμω θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ζημάνσκι, ο οποίο θέλησε να παρέμβει για πέντε λεπτά, γιατί μετά πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσει. Μετά όμω θα ακούσουμε την συνάδελφο Δελβό ούτως ή άλλως. Ο κύριος Ζημάνσκι τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά πρέπει να φύγω ακριβώς στις 11, οπότε έγιναν τόσα πολλά σχόλια που θα ήθελα κάποια να τα, να τα ε, αναπτύξω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα μια προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση προς όλους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, ξεφύγουμε από τη σωστή λογική εδώ. Μην προϋποθέτουμε ότι υπάρχει ένα χρυσό μέσο, μια ε, χρυσή μέση τομή που θα μας επιτρέψει να βρούμε την τέλεια λύση. Δεν υπάρχει μία προσέγγιση που θα ε, δώσει την σωστή συνταγή. Χρειάζονται μια, ένα συνδυασμό μέτρων, ανταγωνιστικότητα, πολιτικές, ε, ποικιλομορφία, πράγματα που θα συνδυαστούν μεταξύ τους. Είναι σαφές αυτό. Θέλουμε όχι να περιορίσουμε τις πολιτικές, αλλά αλληλοσυμπληρωματικές πολιτικές, ε, για να συνδυάσουμε και όλους τους πόρους. Στην Ευρώπη έχουμε συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πυρηνική ενέργεια. Χρειάζεται να γίνει η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια. Χρειάζεται να γίνει η απαραίτητη ανάμειξη, το ενεργειακό μείγμα που έχουμε ε, πει και να δημιουργηθεί μια εύρυθμη ευρωπαϊκή αγορά. Χωρίς αυτό δεν θα επιτύχουμε να βρεθεί μια τοπική πηγή ενέργειας που να λύσει την κατάσταση και όλα τα προβλήματα. Ούτε οι ανανεώσιμε πηγέ μόνο του αρκούν, ούτε το σχιστολιθικό αέριο. Χρειάζεται ένα μείγμα και μάλιστα στι σωστέ δόσει για να πετύχουμε το στόχο μα. Εκπλήσωμε παρόλα αυτά που τόσοι πολλοί συνάδελφοι αναφέρουν την Κίνα ως παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ της πολιτικέ. Η Κίνα είναι η κατεξοχήν χώρα που κάθε εβδομάδα νομίζω κατά μέσο όρο προσθέτει ένα εργοστάσιο το οποίο κινείται με ορυκτά καύσιμα στο οπλοστάσιο εργοστασίων που διαθέτει. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά και φορολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και αυτή τη στιγμή τους στηρίζουν στον προπολογισμό τους. Καλή τους τύχη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλή ενεργειακή τους πολιτική. Δείτε τον αριθμό οχημάτων που κινούνται. Πόσοι οδηγούν στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Όλα λειτουργούν και κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Όχι με ατμό. Αυτό θα ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά τέλος πάντων. Ε, να επικεντρωθούμε στη δική μας την εμπειρία και στο δυναμικό που εμείς έχουμε. Με τις πηγές ενέργειας που ήδη διαθέτουμε. Συμβατικές ή λιθικό αέριο. Συμφωνώ, συμφωνώ, δεν θα αλλάξει το παγκόσμιο σκηνικό από αυτό, αλλά υπάρχουν χώρες που πληρώνουν διπλάσιο τίμημα από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανέφερε η κυρία Χολ, και σε τέτοιε χώρε η ανταγωνιστικότητα μπορεί να τονωθεί. Μιλάμε λοιπόν και για ένα εργαλείο τη αγορά. Δεν θα αλλάξει ολοσχερό το τοπίο, αλλά θα στηρίξει την αγορά. Δεν θέλει η έκθεση λοιπόν να κρίνει, αλλά να συνδυάζει τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε με του πολιτικού μα στόχου. Πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε κατά πόσον τα πολιτικά μα εργαλεία εξυπηρετούν του στόχου που επιδιώκουμε. Μετά από πολλά χρόνια ε, εφαρμογή του πακέτου για τον Ευρώπη του 2020, ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Εάν δούμε λοιπόν τι εισαγωγέ και εξαγωγέ, θα παρατηρήσουμε τι ε, αποκλήσει υπάρχουν. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξαναδούμε την κατάσταση από κάποια απόσταση και να την αποτιμήσουμε. Η κατάσταση προ την ενεργειακή αποδοτικότητα τη ανανεώσιμε πηγέ δεν έχει στρεβλωθεί όπως λέγεται. Αλλά εάν δεν πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, η πολιτική μας τι θα κάνει. Από καιρού καιρών θα ε, προκαλεί νέε εντάσει νέε διαφιλονικίε και αστάθεια. Αστάθεια προ το ρυθμιστικό μας πλαίσιο. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Τα αορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Ωραία είναι αυτή η δήλωση. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία κατά τις πολιτικές μας ε, συναντήσεις ή εκδηλώσει, αλλά απέχει πόρα από την πραγματικότητα. 80% όλων των ενεργειακών, ε, όλη τη ενεργειακή ζήτηση για τα ερχόμενα χρόνια θα καλύπτεται από ορυκτά καύσιμα ακόμα. Κατά εξοχήν από τον ε, άνθρακα. Δεν χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα προτιμούσα να έχουμε αιωλική ενέργεια ή ηλιακή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να μείνουμε σε επαφή με την πραγματικότητα. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε εδώ μονομερή προσέγγιση. Η έκθεση το αντίθετο επιδιώκει να έχουμε πολυμερή προσέγγιση προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Στόχους που να είναι οικονομικά βιώσιμοι αλλά και ενδιαφέροντες για τους εταίρους μας. Όχι μόνο για μας τους ίδιους απομονωμένα. Θα πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε, να τους πείσουμε ότι ο δρόμος μπορεί να μην είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όμως μπορεί να πετύχουμε κάποιες οροπίες ό,τι αφορά τους οικολογικούς μας στόχους και την ενιακή αυτάρκεια. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ τον κύριο Σιμάνσκι. Να κλείσουμε με τις παρεμβάσεις. Κατά πρώτα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στη συνάδελφο Ντελβό. Ο κύριος Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και περισσότερο τόλμη. Και το έκαναν αυτό, νομίζω, οι συνεισηγητέ. Θα μπορούσαν όμω να κάνουν και περισσότερα για την ολοκλήρωση τη ενεργειακή αγορά. Νομίζω αυτό είναι ο τρόπο για να έχουμε την μέγιστη δυνατή χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια από τη μια, από την άλλη όμω να έχουμε ισοτιμία και ίσο κόστο ε, για την τιμή τη ενέργεια για τι εταιρείε και του πολίτε. Ένα παράδειγμα από την Ιταλία, ένα παράδειγμα που είναι τρομακτικό. Οι Ιταλικέ εταιρείε πληρώνουν 130% περισσότερο από τις γαλλικές ή πολωνικές εταιρείε για την τιμή τη ενέργεια. 80% περισσότερο από τις γερμανικές εταιρείε και αν δούμε τι γίνεται με τρίτες χώρε, 400% περισσότερο από ότι οι αμερικανικές εταιρείε. Άρα, τι χρειάζεται. Στην Ευρώπη τουλάχιστον στην Ευρώπη να υπάρχει ίσω ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που ε, ε, λειτουργούν στην ίδια αγορά. Ελεύθερη με αγορά, αλλά που ανήκει στην ίδια ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, βαριές δεσμεύσεις, τις ε, έντονες δεσμεύσεις, είτε για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε για την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στοιχεία που επιβάλλουμε στην, στον κλάδο της ενέργειας, θα πρέπει να προβλέψουμε υποχρεώσεις μεν, αλλά και αποζημιώσεις για εταιρείες που λόγω χάρη λειτουργούν σε τρίτες χώρες και μετά εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κόστος ανταγωνιστικό πληρώνουν πολύ λιγότερο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν ε, ίσω ε, λιγότερε δεσμεύσει ή ε, λιγότερο βάρο ω προ την επίτευξη των στόχων των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την ανταγωνιστικότητά μα και ω προ τον χώρο των επιχειρήσεων. Εντάξει λοιπόν, έχουμε εξαιρετικέ υποσχέσει και δεσμεύσει στην επικρατεία μα στην Ευρώπη. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι άλλοι θα πρέπει να τηρούν του ίδιου κανόνε ή τουλάχιστον να πληρώνουν κανένα δασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρώση, η κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που επανειλημμένως οργανώνεται ε, και στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικότατο. Πράγματι, το κλίμα και η ενέργεια είναι θέματα κέρια σημασίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, το έδειξε και η κρίση αυτό. Ε, κατεπήγει να αλλάξει το μοντέλο μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τη σκοπιά και της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως όλα αυτά να φέρουν κερδοφορία ε, και θέσεις απασχόλησης. Υπ' αυτήν την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο των φιλοδοξιών της και τον ηγετικό της ρόλο την μάχη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Δηλαδή πρέπει να είναι και φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θα πρέπει και να προωθήσει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν ε, μπορεί κανείς να καταλάβει πώς θα στηρίζει ακόμα, ε, θα επιδοτεί τα, τα καύσιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον δεν θα είχε νόημα. Θα πρέπει επίσης να γίνουμε πιο απαιτητικοί ω προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Για να επιτεθεί ασφάλεια και μείωση του κόστους πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση των πηγών τις οποίες ανατρέχουμε. Ακριβώς δηλαδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να διασφαλίσουν το μέλλον μας. Υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να πορευτούμε προς αυτή τη λύση. Ε, λύση προτεραιότητας προασπίζομαι τη λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενεργειακή πολιτική κοινή. Κοινή, ώστε όπως υπόθηκε από αρκετούς συναδέλφους, ώστε να μην Υπάρχουν χώρες που έχουν μία συγκεκριμένη στατικική, άλλη μια διαφορετική. Νομίζω οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ψηλή τιμή για την ενέργεια δεν μπορούν να ανταγωνιστούν εταιρείες που πληρώνουν λιγότερα. Αυτός λοιπόν είναι ένας στόχος που πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο την κυρία Στρέλα και ο κύριος Λίζε έχει ξαναζητήσει το λόγο. τρεις διευκρινήσεις για να αποφύγω οποιαδήποτε παρανόηση. Ο κύριος Λάγκεν είπε κάτι σημαντικό, το οποίο επανέλαβε λίγο πολύ και η κυρία Εστρέλα. Ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών δεν έχουμε αρκετή συνεννόηση και εξισορρόπηση και σωστό είναι που το λέει και η κυρία Ντελβό στο κείμενό της. Αυτή η έλλειψη συντονισμού για τις ανανεώσιμες ενέργειες αποτελεί πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε δίκτυα, να επενδύσουμε σε τρόπους αποθήκευσης των ενεργειών, επίσης καλύτερα το demand management, αν θέλουμε να συνεργαστούμε διαμεθοριακά, που είναι απαραίτητο. Χωρίς αυτό όμως να έρχεται σε αντίθεση με δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Εάν δεν συνεχιστεί η επέκταση των ανανεώσιμων ενεργειών, δεν θα έχουμε και τίποτα να εξισορροπήσουμε ή να συντονίσουμε. Το μεγάλο αδύναμο σημείο του μέχρι τώρα πακέτου κλίματος και ενέργειας είναι ότι δεν έχουμε βάλει δεσμευτικό στόχο για την αποδοτικότητα της ενέργειας και ότι τώρα εκ των υστέρων ερχόμαστε να φτιάξουμε μια οδηγία η οποία θα βέβαια συνεπιφέρει προβλήματα ιδίως στο εμπόριο εκπομπών. Βέβαια τα πράγματα στη ζωή δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι σε ολόκληρο τον κόσμο όλοι θα μιμηθούν τις πολιτικές μας. Αυτά όμως που λένε οι κύριοι Σιμάνσκι και άλλοι ότι δεν γίνεται τίποτε ανά τον κόσμο, αυτό σίγουρα είναι λάθος. Με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος βρεθήκαμε στην Ουάσιγκτον και ακούσαμε ότι για παράδειγμα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα οι τιμές που εγκρίθηκαν ήδη στις ΗΠΑ και μάλιστα μακροπρόθεσμα είναι ακόμα αυστηρότερες από αυτές τις οποίες διαπραγματευόμαστε εμείς τώρα. Ο δε πρόεδρος Ομπάμα προωθεί νομοσχέδιο που λέει Διακοπή από τον κύριο Λάγκεν χωρίς μικρόφωνο. Βεβαίως δεν μπορεί να κάνει κανείς συγκρίσεις 100% αλλά ως παράδειγμα το λέω ότι εκεί στην Αμερική δηλαδή υπάρχουν πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος. Ασφαλώς και υπάρχουν εξαιρέσεις και εκεί και αλλού. Τελευταίο σχόλιο υπάρχει νομοθετική πρόταση. Με διακόπτει ο κύριος Λάγκεν κυρία Πρόεδρε Η Ελίζα είναι η δεύτερη σας παρέμβαση. Να ολοκληρώσω τη φράση μου κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει πρόταση που μπορεί να εγκριθεί χωρίς την συμβολή του Κογκρέσου για οριακές τιμές για εργοστάσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο από ορυκτά καύσιμα. Αυτέ οι τιμέ είναι πολύ αυστηρότερε από ό,τι θα μπορούσαμε καν να διανοηθούμε στην Ευρώπη. Άρα δεν ισχύει διόλου το ότι δίθεν εμεί μονάχα σε όλο τον κόσμο κάνουμε προστασία του κλίματος. Ευχαριστώ, αλλά σα θυμίζω ότι καλό είναι να σεβόμαστε το χρόνο ομιλία. Είναι μία από τι βασικέ προποθέσει για να έχουμε μια ειρηνική συζήτηση. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Φεργότε, υπεύθυνο για την οικονομική αποτίμηση τη Γενικής Διεύθυνσης για το Κλίμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συνεισηγητές για την έκθεση αυτή που είναι πολύ σημαντική για μας. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα πακέτο σε σχέση με το 2030 που θα παρουσιάσει σύντομα στις αρχές της επόμενης χρονιάς κατά πάσα πιθανότητα. Να απαντήσω σε κάποια από και να σχολιάσω κάποια από αυτά που ακούσαμε. Πολλοί ακούσαμε για την ισορροπία ανάμεσα στον ενεργειακό εφοδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του κλίματος. Όντως η ισορροπία αυτή είναι στο κέντρο της συζήτησης, γι' αυτό και εμείς θέλουμε ένα συντονισμένο πλαίσιο που να ασχολείται και με τα τρία. Και ένα από τα θέματα που ανέφεραν κάποιοι και υπάρχει και στην έκθεση, είναι για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 5 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια 3,2% του ΕΠ και το διπλάσιο από ό,τι είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια, η αύξηση στις τιμές δηλαδή. Κάτι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά μας. Άρα χρειάζεται ισορροπία και συνέργειες ανάμεσα στις διάφορες πτυχές των πολιτικών μας ενέργειας και κλίματος. Έχουμε πολλά για την ενεργειακή απόδοση, για την καινοτομία, τα οποία ήδη αρχίζουν να δημιουργούν συνέργειες. Δεύτερον, ο κύριος Γιμάσκι μίλησε πολύ για δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όσον αφορά το κλίμα αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το είπανε και πολλοί άλλοι. Αυτή τη βδομάδα αρχίζει το νέο κοπ που αποτελεί άλλον έναν ακρογωνιαίο λίθο σε σχέση με το 2015 που αποφασίσαμε να πετύχουμε συνολική λύση για την περίοδο μετά το 2020. Το ενθαρρυντικό είναι ότι στην τελευταία συνάντηση και η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι θα προτείνουν σχέδια για το τι θα κάνουν δηλαδή μετά το κόψτο στο Παρίσι του 2015, τι θα κάνουν μετά το 2020. Άρα ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιριών, εφόσον οι δύο που εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακο, θα μας πούνε σε δύο χρόνια, ενάμιση, τι τελικά θα κάνουν. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για τις προσπάθειες που κάνουν οι άλλοι. Έχουμε το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Επιτροπής που κάθε χρόνο δημοσιεύει έκθεση για τις παγκόσμιες εκπομπές και κάθε χρόνο η έκθεση αυτή είναι μια κακή είδηση. Κάθε χρόνο λέει ότι έχουμε αύξηση των εκπομπών και μάλιστα πολύ γρήγορη κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό σε σχέση με το στόχο μας τους δύο βαθμούς ανώτατη αύξηση στο κλίμα. Τώρα όμως βλέπουμε ξαφνικά ότι υπάρχει μια διαφορά. Για πρώτη φορά ρητά η έκθεση αυτή δείχνει ότι τα μέτρα που παίρνουν οι αναπτυσσόμενες επίσης χώρες αποδίδουν η Κίνα για παράδειγμα. Αυτή η έκθεση λοιπόν το καταδεικνύει. Τέλος, για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων και το μη σύστημα είναι σημαντικό να ξέρουμε εδώ ότι η διαβούλευση που έγινε μετά την πράσινη βίβλο έδειξε ότι υπάρχει συνένεση για το ότι το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπή είναι το πιο βασικό σύστημα ω κίνητρο για την μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό πράγματι να έχουμε κοινή στάση στην Ευρώπη και όχι κατακαιρματισμό. Διάσταση απόψεων εμποδίζει την εφαρμογή της πολιτικής μας άρα αυξάνει το κόστος. Τέλος, πολλοί ομιλητές, η κυρία Χολ μεταξύ άλλων, είπε ότι είναι σημαντικός και ο τομέας εκτός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Μεταφορές, κτίρια, εξοικονόμηση, εφοδιασμός, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στους τομείς αυτούς πολύ. Είναι καλό λοιπόν που η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι τομείς αυτοί έχουν μεγάλη σημασία σχετικά με την τελική προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Χορτόφερ, υπεύθυνο των κλιματικών πολιτικών της Γενικής Διεθνής, υπεύθυνο της Γενικής Διεθνής Ενέργειας. Και εμείς της Γενικής Διεθνής Ενέργειας ευχαριστούμε τους δύο εισηγητάς και θεωρούμε την έκθεση υπό την μορφή που έχει επιβληθεί ότι θέτει σωστά τα θέματα για την ενεργειακή πολιτική. Βεβαίως πρώτα αποδοτικότητα της ενέργειας για μας είναι σημαντικό να παραμείνει από τα πιο σημαντικά ορόσημα. Προβλέπουμε εμείς έκθεση για το 2014 στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας Άρα στην έκθεσή μας για το 2030 θα αναφερθούμε στην αποδοτικότητα της ενέργειας. Πέραν αυτού όμως θα τονίσουμε επίσης ότι το 2014 έρχεται η οδηγία για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Καλύπτονται λοιπόν αυτά και τα δύο. Ανανεώσιμες ενέργειες εξακολουθεί να παραμένει no regret option, όπως είπαμε και στο οδικό, στον οδικό χάρτη. Είναι σωστό ότι σε διάφορες χώρες μέλη υπάρχουν διάφορα μέτρα για αναδρομικές περικοπές των επιδοτήσεων. Τα βλέπουμε όμως αυτά και σε ορίζοντα 2030 και θεωρούμε σημαντικό τον ρόλο των ανανεώσιμων ενεργειών, διότι άλλωστε πρόκειται για δικό μας πόρο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Τονίζονται στην έκθεση, έκθεση και η υποδομή, που και για μας είναι σημαντική, σημαντικότατος τομέας για την ενέργεια. Οι χώρες μέλη πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο. Εμείς Κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι ο στόχος του 2014 με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και τη συνέχιση παραμένουν σημαντικά. Ορισμένοι βουλευτές έφυξαν το θέμα των τιμών της ενέργειας. Στην έκθεση για το 2030 θα αναλύσουμε τα σχετικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε στο impact assessment με βάση διάφορα σενάρια και με μέτρα αποδοτικότητας τη ενέργεια και εκεί θα φροντίσουμε να περιληφθεί η ανάλυση των τιμών. Εκτός αυτού όμως, τον Μάιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να προβεί σε λεπτομερή ανάλυση του κόστους και των τιμών της ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε σύγκριση με τους μεγάλους ανταγωνιστέ μα. Αυτά θα τα πράξει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή μέχρι τέλου του έτου ή αρχών του επομένου Έτου. Εδώ κρύβεται ένα σημαντικός παράγοντας για την αύξηση των τιμών που είναι τα ορυκτά καύσιμα. Είναι σαφές αυτό. Θα αναλύσουμε βεβαίως επίσης και ποιες είναι οι άλλες συνιστώσεις. Ποιος είναι ο ρόλος των ανανεώσιμων ενεργειών. Επίσης της φορολόγησης των καυσίμων. Και αυτά θα τα περιλάβουμε ως συμπληρωματικά δεδομένα για το 2030. Από την άποψη της ενεργειακής πολιτικής, νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά που θέλω να σχολιάσω. Όπως είπα, συντάσσουμε το έγγραφο τώρα για τον Γενάρη και γι' αυτό η σημερινή συζήτηση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και η επομένη που θα κάνετε, είναι πολύ σημαντικές για μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τα τόσο ενδιαφέροντα σχόλιά σας, τα οποία βέβαια με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ, είναι κάπως απλοϊκό να πούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλη αυτή την προβληματική με ένα μόνο στόχο. Να κάνω όμως και μια διευκρίνηση, αναφέρθηκε στο θάρρος ο κύριος Ρώση και άλλοι ίσως να έχουν δίκιο. Μερικές φορές λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία και διευκρινήσεις στο κείμενο αυτό. Το κείμενο όμως αυτό αποτελεί καρπό συνένεσης μεταξύ δύο συνεισηγητών. Και τα πιο συγκεκριμένα θα αντέχουμε με τις τροπολογίες. Θα απαντήσω τώρα στα σχόλια ορισμένων, οι οποίοι βέβαια έφυγαν, αλλά δεν πειράζει. Κύριε Ιλσκοκ, αναρωτήθηκε για την ανταγωνιστικότητα και ότι βάζουμε σε αντιπαράθεση την ανταγωνιστικότητα με την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, όχι λοιπόν. Εγώ αυτό θέλω να το διευκρινίσω ότι για μένα είναι ξεκάθαρο πως η ενεργειακή απόδοση και η ανταγωνιστικότητα πάνε μαζί υπό τον όρο όμως να υπάρχει σωστή πλαισίωση να δούμε τη σχέση κόστους και δαπάνης και να δούμε και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Και όταν μιλάμε για απόδοση, εδώ θέλω να επιμείνω και πάλι στην ενεργειακή απόδοση. Αποτελεί το νέο ακρογωνιαίο λίθο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και υπογραμμίζει την δυνατότητα να προχωρήσουμε, όπω είπε και η κυρία Χόλ πριν από λίγο, να προχωρήσουμε και στου τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπή αερίων, Μεταφορέ, κτίρια. Πράγματι πρέπει να τονίσουμε και αυτόν τον τομέα. Και τον κύριο Λίζε και τις ανανεώσιμες πηγές. Υπενθυμίζω ότι γίνεται συντονισμός. Εγώ τουλάχιστον ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Γιατί στον τομέα των επιδοτήσεων στις ανανεώσιμες πρέπει να είναι πιο στοχοθετημένη η δράση μας και ενδεχομένως να στρέψουμε τις επιδοτήσεις προς άλλες ανανεώσιμες πηγές που δεν έχουν οριμάσει ακόμα αρκετά και να τις βγάλουμε τις επιδοτήσεις αυτές από τις ε, όριμες ανανεώσιμες πηγές. Για άλλους οι οποίοι δεν είναι πια εδώ θέλω να σας πω ναι και τις επιδοτήσεις στα ορυκτά πρέπει να ξαναδούμε για να υπάρχει συνοχή. Έρχομαι τώρα στο θέμα της τιμής. Πάλι εδώ ένα πλοϊκό να λέμε ότι φταίνε ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχει και το θέμα των φόρων που αποφασίζονται στα κράτη-μέλη. Άκουσα από την Επιτροπή ότι ίσως να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση για το κόστος σε εθνικό επίπεδο στις 28 χώρες. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί, αλλά ρεαλιστές όσον αφορά τη σύνθεση το μείγμα των τιμών και να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για το μείγμα αυτό. Δεν είναι μόνο το κόστος, πρέπει να ξέρουμε πώς φτάνουμε σε αυτό το κόστος. Και είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες να υπάρχει διαφάνεια. Ναι, να μιζάρουμε στην έρευνα, την καινοτομία. Όντως αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να κρατηθούν καλύτερα μέσα στον ανταγωνισμό. Κύριε Στρέλ, έχετε δίκιο, πρέπει να επιμείνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έχω ήδη πει. Είναι παράδεκτο μια χώρα να αποφασίζει από μόνη της να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα. Χωρίς καν να ενημερώσει, για παράδειγμα, τις γείτονες χώρες. Για μένα είναι παράδεκτο κάτι τέτοιο. Εάν θέλουμε να πάμε προς μια αγορά χωρίς πυρηνικά, τότε θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική επικοινωνίας μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί συνεργασία μεταξύ χωρών μελών. Χρειαζόμαστε διάφορα μέσα, το είπε και ο κύριος Σιμάνσκι πριν από λίγο και γι' αυτό εξάλλου και εμείς θέλουμε ένα πιο ευρύ ενεργειακό μείγμα. Γιατί θέλουμε οι τεχνολογίες να είναι στραμμένες στο μέλλον. Γιατί η απασχόληση είναι κεφαλαιόδου σημασία επίσης. Το είπα και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε τρεις δεσμευτικούς στόχους, αλλά να είναι καλά πλαισιωμένοι. Να πάρουμε μαθήματα από το πακέτο που είχαμε μέχρι τώρα. Φιλοδοξίες ναι, αλλά και ρεαλισμός. Ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Δεν θέλω να την ξανανοίξουμε. Κυρία Ζέμπερ. Εδώ λέει στο δικό μου το χαρτί 12.30 τέλος. Τώρα είναι 11 και 20. Σας είπα όμως στην αρχή, δύο ώρες για τη συζήτηση. Λάθος της γραμματείας. Το είπα ευθύς εξ αρχής. Δύο ώρο. Δεν μου αρέσει να δίνω υποσχέσεις κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι σημαντική η συζήτηση και είμαστε μαζί με την ε, Επιτροπή Βιομηχανίας. Μιλεί και η πρόεδρος με το μικρόφωνο ανοιχτό. Θα είχα προτιμήσει όμως να ζητήσετε το λόγο πριν την ολοκλήρωση και πριν την Επιτροπή. Ε, περίμενα, εν πάση περιπτώσει, έχω μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Έχουμε την ψηφοφορία στις 9 πρώτου. Έγκριση της ε, εκθέσεως στην Ολομέλεια τον Φεβρουάριο. Γιατί δεν περιμένει η Κομισιόν μέχρι ότου εγκρίνουμε την έκθεση αυτή εδώ στο Κοινοβουλίο. Μήπως δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνει το Κοινοβούλιο. Επιτροπή, σα τέθηκε ένα ερώτημα. Ποιος θα απαντήσει. Ή ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο το Μάιο, να παρακολουθήσει το πώ. ποια ήταν η απήχηση τη πράσινη Βίβλου, Έως τον Νοέμβριο φέτος ε, με, την, ε, με τη Σύνοδο του Συμβουλίου. Νομίζω ότι το Γενάρη κάτι πρέπει να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αργότερα θα ήταν πολύ δύσκολο εν ώψη του Συμβουλίου του Μαρτίου. Αλλά προηγουμένως και η Διεπιτροπή μας και ε, ο πρόεδρος μας ευχαρίστως να σας παρακολουθήσει. Το πρώτο βήμα είναι αυτό Τη η συζήτηση και η ψηφορία που θα γίνει στις αρχές Ιανουαρίου. Νομίζω ότι αν τον Ιανουάριο υπάρξει κάποια πρόοδος, υπάρχει κάποια εξέλιξη, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να ληφθεί πλήρως υπόψη. Ευχαριστώ. Νομίζω η παρέμβαση του κ. Ζέμπερ ήταν ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά. Να ζητήσουμε λοιπόν από τον Επίτροπο να μας περιμένει. Χρόνος υπάρχει. Ε, συνάδελφε Γκρότα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρήκα πολύ καλή την συζήτηση και απευθύνομαι στην Κομισιόν τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Καλά θα κάνετε να λάβετε υπόψη τα όσα συζητεί το Κοινοβούλιο, διότι στο κάτω της γραφής εμείς είμαστε οι νομοθέτες. Χωρίς εμά, εμάς δεν περνάει τίποτα. Εμείς θα διαθέσουμε στους αυτές μας τον απαραίτητο χρόνο, διότι θα είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί το θέμα αυτό, που άλλωστε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλαγή του κλίματος, πολιτική της ενέργειας. Γνωρίζουμε ότι αυτά διέπουν τις σκέψεις και τις πράξεις μας και όλες βέβαια οι πτυχές της οικονομίας. Εάν κανείς κάνει το συνολικό λογαριασμό, αυτά τα πράγματα πρέπει να φωτιστούν πολύ περισσότερο. Διότι ένας τομέας της οικονομίας ακόμα δεν λήφθηκε παλκώς υπόψη. Ιδίως δηλαδή η, ο κλάδος των ασφαλίσεων. Τι θα σημάνει αν τα πράγματα συνεχιστούν όπως μέχρι τώρα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Τι θα κάνει ο ασφαλιστικός κλάδος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστή η έκθεση, έχει σωστό προσανατολισμό. Πιστεύω ότι ακόμα ορισμένες χώρες μέλη δεν έχουν κατανοήσει ότι εδώ η Ένωση είναι αρμόδια για την ενέργεια από 1η πρώτου του 2009. Το energy mix το κάνουν οι χώρες, αυτό είναι σωστό, αλλά πρέπει να γίνει καλύτερη εναρμόνιση. Ο καθένας μαγειρεύει στην κουζίνα του εκεί πέρα, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρξει ένας κεντρικός συντονισμός. Στοιχεία, δεδομένα τα οποία έχουμε κοινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ρυθμιστούν κοινά, γιατί αυτό είναι και οικονομικά σωστό και οικολογικά. Καλά περάσαμε μαζί με τους συναδέλφους της Ήτρε, έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε σε αυτή τη συνεργασία. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η συνεδρίαση και πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή δείχνουν πνεύμα συμβιβασμού. Ευχαριστούμε συνάδελφε Γκρότ. Νομίζω θα λύσουμε των προτέρων όλα αυτά τα προβλήματα που δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε πάντοτε εκ των υστέρων. Να θυμίσω ότι η διορία για τις ε, τροπολογίες είναι στις 12 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Το σχέδιο έκθεσης θα διατεθεί στο, σύστημα από τις τέσσερις για να μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες και θα πρέπει να αποστείλετε με φάξ όλες τις αιτήσεις σας προς την γραμματεία. Στη φάση αυτή σας ευχαριστώ όλους. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι η επόμενη συνεδρίαση, κοινή συνεδρίαση ΕΝΒΙ ΙΤΡΕ προβλέπεται για τις 2 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Καλή σας ημέρα και καλή δουλειά.